Varmt välkomna till dagens utskottsmöte för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Ερχόμαστε λοιπόν στην ημερήσια διάταξη και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ε, σας ρωτήσω κατά πόσο συμφωνείτε συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη, επιθυμεί κάποιος να αλλάξει κάτι σε αυτήν. Ε, πρόκειται για την ε, βελτίωση ε, της ασφάλειας και της θέσης της εργασίας. Η κυρία Στρέλα είναι η η για το θέμα αυτό, η οποία αύριο, λίγο μετά τις 11, είναι αναγκασμένη να φύγει. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω το θέμα αυτό να το εξετάσουμε αύριο αμέσως μετά τη συζήτηση για τα θέματα 11 και 12. Το 10 λοιπόν θα είναι αύριο το τελευταίο σημείο της μερικής διάταξης. Συμφωνείτε επ' αυτού. Πολύ ωραία λοιπόν. Ε, άλλαξε κατά τη μόνο η ημερήσια διάταξη. Πάμε στο επόμενο σημείο που είναι η έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 29-30 Σεπτεμβρίου 2009. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις ε, μέχρι το τέλος της ε, σημερινής συνεδρίασης θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Σημείο 4. Ανακοινώσεις της Προέδρου Εδώ έχω... Εδώ έχω λίγα πράγματα να σας πω, αλλά παρακαλώ να τα σημειώσετε. Η επόμενη συνάντησή μας θα λάβει χώρα τον ε, Ιανουάριο και εκεί θα έχουμε το απόγευμα ψηφοφορία στις 25 Ιανουαρίου. 25 Ιανουαρίου λοιπόν θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία γύρω στις 4 ε, και 4. Κατόπιν. 26 Ιανουαρίου και για την 26η Ιανουαρίου έχει προβλεφθεί συνεδρίαση, όμως ε, πρέπει να αλλάξουμε λιγάκι αυτήν την ημέρα, γιατί στις 26 ε, Ιανουαρίου τελικά αποφασίστηκε να είναι η μέρα Ολομέλειας, όπου θα ψηφίσουμε για τους νέους επιτρόπους. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν την ίδια εβδομάδα έχουμε κάποια άλλη μέρα για να συνεδριάσουμε και μόλις ενημερωθούμε τελικά τι θα γίνει με τους ε, διερμηνείς ε, και με τις αίθουσες ε, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν για να σας πούμε ποια ακριβώς η μέρα θα λάβει, ε, ποια ώρα πιο συγκεκριμένα ή και ποια μέρα ναι, θα λάβει η χώρα αυτή η συνεδρίαση, γιατί σας είπα 26 Ιανουαρίου δυστυχώ είναι αδύνατον. Παρακαλώ λοιπόν να συγκρατήσετε αυτές τις ε, πληροφορίες για την επόμενη συνεδρίασή μας τον Ιανουάριο. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι το υπαριθμόν 5. Πρόκειται για την απαλλαγή του 2008. Γενικός Προϋπολογισμός, ε, τμήμα 3, Επιτροπή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμών μας ενημέρωσε για τη διαδικασία που αφορά στην απαλλαγή του 2008. Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του 2010 πρέπει να τοποθετηθούν όλες οι επιτροπές. Το χρονικό διάστημα είναι μικρό, τουλάχιστον έτσι το βλέπουμε εμείς, όμως ε, εμείς ε, αποφασίσαμε να γνωμοδοτήσουμε η κυρία Μπάουα ανέλαβε τη γνωμοδότηση εκ μέρους της Επιτροπής μας και γι' αυτό λοιπόν το λόγο προτείνω να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτή τη γνωμοδότηση. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στην κυρία Μπάουα για να μας ενημερώσει σχετικά με το θέμα αυτό. Παρακαλώ κυρία Μπάουα, έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη. Δεν ξέρω ε, κατά πόσον ε, υπάρχει διερμηνία σε όλες τις γλώσσες. Εμείς ε, συντάξαμε τη γνωμοδότηση στα αγγλικά γιατί δεν είχαμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Πέτε από τη Γραμματεία, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να εξετάσει κανείς το θέμα αυτό, κυρίως χωρίς υποστήριξη. Αλλά εμείς, εν πάση περιπτώσει, ήμασταν τυχεροί, δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα, είχαμε την αμέριστη υποστήριξη της ε, γραμματείας. Στην Επιτροπή, λοιπόν, εκπονήθηκε μία μελέτη, Gender Budgeting είναι η επικεφαλίδα, η μελέτη αυτή υπάρχει και θα ήθελα να σας επισημάνω και κάτι άλλο. Το όνομα αυτού του Ινστιτούτου για τα δύο φύλλα, του Gender Institute, ε, δεν εμφανίζεται γιατί ε, είναι σχετικά ε, πρόσφατη η σύστασή του και γι' αυτό δεν έχει και προπολογισμό το Ινστιτούτο. Ως εκ τούτου δεν έχει και όνομα. Κάτι άλλο που θέλω να επισημάνω. Δεν έχουμε αρκετά στοιχεία στη διάθεσή μας ε, που να μπορούν να μας ενημερώσουν ε, καλύτερα για την ε, κατανομή των δύο φύλων. Θελήσαμε λοιπόν σε αυτή τη γνωμοδότηση να συντάξουμε κάποια στατιστικά δεδομένα τα οποία αναφέρουμε στην εκθεσή μας και με μεγάλη ανυπομονωσία περιμένω την τοποθέτηση των συναδέλφων. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπάουερ. Και σας ευχαριστώ που επισημάνατε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την έλλειψη μεταφράσεων στις άλλες γλώσσες. Μόλις σήμερα λάβαμε το έγγραφο και μάλιστα μόνο στα αγγλικά. Θα μεταφραστεί όμως και στις υπόλοιπες γλώσσες. Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου περίπου πριν λήξει δηλαδή η προθεσμία για την κατάθεση των απολογιών. Μπορούμε να προβούμε σε μια ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό της απαλλαγής ε, του προϋπολογισμού 2008. Eh, Κυρία Μπάουερ, ε, συντάξετε μια καταπληκτική γλωμοδότηση, γιατί φαίνεται ότι κανένας δεν έχει αντιρρήσεις, παρατηρήσεις. Συγχαρητήρια θερμά κυρία Μπάουερ. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα τώρα. Η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών λήγει στις 15 Δεκεμβρίου το μεσημέρι. Ευελπιστούμε ότι θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 25 Ιανουαρίου. Τη Δευτέρα το απόγευμα δηλαδή, 25 Ιανουαρίου, τότε προβλέπεται η ψηφοφορία της έκθεσης αυτής. και στις 22 ε, και 23 Μαρτίου θα ψηφίσει η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο και να περάσουμε στο επόμενο. Την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε χρόνο και ύστερα από αίτημα των θεσμικών οργάνων yes. καταρτίζεται έκθεση για την πρόοδο που σημειώνουμε στα θέματα ισότητας των δύο φύλων και εξετάζονται οι προκλήσεις ε, για το μέλλον και οι προτεραιότητές μας. Μάλιστα υπάρχει και η δυνατότητα να συντάξουμε έκθεση ίδιες πρωτοβουλίας. Και μάλιστα αυτή η έκθεση δεν εμπίπτει στον πεπερασμένο αριθμό εκθέσεων ίδιας πρωτοβουλίας που έχουμε. Ε, μάλιστα, αν, το, αν την εκπονήσουμε αυτή την έκθεση, θα περάσει στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου. Ή του Φεβρουαρίου, συγγνώμη. Η συγκητής τη ε, έκθεσης αυτής είναι ο κύριο Ταραμπέλα, στον οποίο και θα δώσω το λόγο. για να μας ενημερώσει για το έργο που έχει γίνει μέχρι τώρα και τι γίνεται με την ισότητα των δύο φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2009. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι, να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθεια την οποία έκανε, ισόρροπη, σωστά διατυπωμένη. Να ευχαριστήσω επίσης ε, τα μέλη της Επιτροπής και για τη διαθεσιμότητά τους. Δεν θα ήθελα να επανάλθω στις λεπτομέρειες. Θα ήθελα να συγκεντρώσω την προσοχή μου σε 7 σημεία τα οποία θεωρώ ότι είναι πιο χρήσιμα. Πρώτον, σχετικά με την οικονομική κρίση. Απεδείχθη ότι η κρίση μπορεί να θίξει σε μία πρώτη φάση και τους άνδρες γιατί υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στις λεγόμενες θέσεις εργασίας, χαλιβουργία κτλ. Βαριά βιομηχανία. Αλλά υπάρχουν και άλλες συνέπειες που ακολουθούν σε μία δεύτερη φάση στις δημόσιες υπηρεσίες και στις κοινωνικές υπηρεσίες όπου εκεί υπάρχει πλειοψηφία γυναικών εργαζομένων. Και γι' αυτό ακριβώς ζήτησα συγκεκριμένες στατιστικές ε, για τις ε, διακρίσεις που κάνει σε εισαγωγικά η κρίση για τους άνδρες και τις γυναίκες και μια ανάλυση επιπτώσεων ανάλογα με το φύλλο πριν προωθήσει κανείς μια δημοσιονομική πολιτική λιτότητα έτσι ώστε οι γυναίκες να μην θίγονται δυσανάλογα Τώρα, για τον χώρο της εργασίας. Εδώ βλέπουμε ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι 59,1 για το 2008. Πλησιάζουμε τους στόχους της Λισαβόνας, αλλά υπάρχουν διαφορές, 25% στη Μάλτα και 57% σχεδόν το διπλό στη Δανία. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να εφαρμόσουν σωστά τις οδηγίες τα κράτη-μέλη. Είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες πλειοψηφούν στις πανεπιστημιακές σπουδέ, στις νομικές σπουδέ, στις εκπαιδευτικές σπουδέ. Έχουν το 58% των τίτλων των πανεπιστημιακών πλέον οι γυναίκες. Και η κορονίδα είναι ότι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις βέβαια εξακολουθούν να μην έχουν κατευθυντήριες θέσεις, διοικητικές θέσεις υψηλού επίπεδου παρά δηλαδή τις εξελίξεις αυτές στον τομέα των διπλωμάτων των ανωτάτων σχολών παραμένουν οι γυναίκες στις ανώτατες θέσεις στο 30%. Σε επίπεδο αμοιβών, διαφορά 17,54%. Ένα βελγικό συνδικάτο που ονομάζονται Γενική Συνομοσπονδία Βελγίου, FZTB, κάνει μία μελέτη και φτάνει στο 25%, λαμβάνοντας υπόψη και το ποσοστό της επιμέρους απασχόλησης που αφορά περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άνδρες. Το 17% είναι η ελάχιστη διαφορά στατιστικά και μπορεί να είναι και πολύ περισσότερη. Έχει σημασία λοιπόν να ζητήσουμε την πραγματική εφαρμογή από τα κράτη-μέλη της συγκεκριμένης οδηγίας που αφορά την ισότητα αντιμετώπισης ανδρών γυναικών στην απασχόληση και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να προωθήσουν την βασική αρχή ίση εργασία, ίση απασχόληση. Τρίτο θέμα, σεξιστικά στερεότυπα. Και οι γυναίκες και οι άνδρες υποφέρουν από τέτοιου είδους στερεότυπα στην επαγγελματική τους και ιδιωτική ζωή. Η κοινωνία δεν θα μπορέσει να εξελιχθεί παρά μόνο όταν ξεπεραστούν οι δυσκολίες αυτές και όταν ο καθένας μπορεί να επιλέξει τη δουλειά που θέλει να κάνει ανάλογα, ανεξάρτητα μάλλον από το φίλο του. Ε, μια ιστοριούλα όταν ήμουνα υπουργό υπεύθυνο για την κατάρτιση και κάποια στιγμή μου επετέθη μια γυναίκα η οποία ήθελε να γίνει οδηγός σχολικού λοφορείου. Έλειπαν θέσει. αλλά παρόλα αυτά είχε πέσει θύμα σεξισμού, όχι από πλευρά των υπολείπων 39 υποψηφίων που ήταν άνδρες, αλλά από πλευρά ε, του καθηγητή που τους είχε πει ότι δεν είναι γυναικεία δουλειά, ότι πρέπει να αλλάξει, να γίνει κομμότρια κτλ. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και όταν ψηφίζουμε νόμους, όταν ψηφίζουμε οδηγίες, παραμένουν δυστυχώς αντιλήψεις και συμπεριφορές επιτόπου οι οποίες είναι αρνητικές. Πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης στα σχολεία, στους χώρους εργασίας για να καταπολεμηθούν αυτά τα στερεότυπα. Και εδώ ίσως να πω και κάτι πρωτότυπο, να υπογραμμίσω ε, τον ρόλο των ανδρών στην ίση κατανομή των οικογενειακών βαρών. Δεν είναι σπάνιο και δεν πρέπει να είναι σπάνιο ε, να, να βγαίνει ένας άνδρας και να αλλάζει τις πάνες του μωρού του. Εμένα μου έχει συμβεί αυτό, τώρα δεν μου συμβαίνει πια γιατί το παιδί μου είναι 4 ετών, αλλά εν πάση περιπτώσει. 35% είναι οι γυναίκες στο κοινοβούλιο, 32% στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Ίσως ε, ο δημόσιος χώρος, η δημόσια ζωή να δίνει ένα παράδειγμα. Το 41% των προέδρων είναι γυναίκες, 42,8% είναι αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους κοσμήτορες, δεν ξέρω αν είσαστε πλειοψηφία οι γυναίκες στους κοσμήτορες. Τώρα είσαστε το 1 τρίτο. Εντάξει, δεν είναι και τόσο κακό. Φυσικά είσαστε ένα τρίτο, αλλά υψηλή ποιότητα. Η κυρία Λούλινγκ είμαι πάντα πεπισμένο ότι αξίζει για δύο. Υπάρχουν λοιπόν βήματα προόδου, σημαντικά, αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλα. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακολουθήσει, ε, ξέρετε, ε, την στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να υπάρχει ένα τρίτο τουλάχιστον γυναικών στις διοικητικές θέσεις ανώτερες. Το πέμπτο σημείο είναι η βία εις βάρος των γυναικών. Αρμοδιότητα περισσότερο της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών. Αλλά ίσως το αρχικό κείμενο αυτό που ζητά για την καθιέρωση ε, μιας ημέρας για εναντίον της ε, βίας εις βάρος των γυναικών. Ίσως θα πρέπει να υπάρξει μια χρονιά για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών. Για να μπορέσουμε να πάρουμε πολύ συγκεκριμένα και εφαρμοστέα μέτρα. Το έκτο είναι οι μετανάστριες. Γιατί, γιατί το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι ένα φαινόμενο το οποίο αυξάνεται συνεχώς, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι δύσκολο να ανακόψει κανείς και στα πλαίσια ακριβώς αυτού του φαινομένου οι γυναίκες περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν νιώθουν μια κάποια εκρίζωση, νιώθουν θύματα διάκρισης ακριβώς και λόγω φύλου και λόγω του καθεστώτος ε, της μετανάστριας. Πολλές φορές ε, θα μπορούσαν να ασχοληθούν με συγκεκριμένες ειδικευμένε θέσεις απασχόλησης αλλά δεν τους δίνεται η ευκαιρία. Ζητάμε λοιπόν από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια καλύτερη προστασία των μεταναστριών και μια προσπάθεια υποβοήθησης της ενσωμάτωσής τους. Να μην παραλείψω να ασχοληθώ και με το πρόβλημα των γενετησίων δικαιωμάτων. Οι γυναίκες θα πρέπει να διαθέτουν το σώμα τους όπως το επιθυμούν αυτή είναι μια αρχή που πρέπει να υπερασπιστούμε, γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε μέτρα για να υπάρχει βελτίωση της ε, πρόσβασης των γυναικών στις υπηρεσίες υγείας και στις υπηρεσίες ε, γενικά που ασχολούνται με την σεξουαλική ζωή των ε, ασθενών, των ανθρώπων. Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι προφανώς και περιμένω τα σχόλιά σας με πολύ ενδιαφέρον και να σημειώσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών, Πρόεδρε, είναι η Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 12η Μεσημβρινή. Σας ευχαριστούμε κύριε Ταραμπέλα. Θα ήθελα να συζητήσουμε αυτή την έκθεση. Πρώτα απ' όλα όμως να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Ταραμπέλα για την πολύ ενδιαφέρουσα επισκόπηση που μας έκανε το του τους, καθώς ε, και τα 7 σημεία στα οποία συνόψισε την έκθεσή του. Νομίζω ότι αυτές είναι και οι βασικές προτεραιότητες του κειμένου και περιμέναμε ανυπομονησία της απόψης και των συναδέλφων για αυτά τα 7 θέματα. Ε, φυσικά, ίσως έχετε και άλλες προτάσεις για προτεραιότητες που κατά τη γνώμη σας καλό θα ήταν να συμπεριληφθούν στην έκθεση. Έχω σημείωση του κατάλογο μιλητών της Σόφη Ιντφελτ και μετά την Ήλτα ε, Φιγκερέντο, την κυρία Λούλινγκ, την κυρία Έρνστ. Πρώτα, όπως είπα, δίνω το λόγο στη Σόφη Ιντφελτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή μας για την καταπληκτική του έκθεση. Και η ομάδα μου σίγουρα θα υποστηρίξει τις αδερές γραμμές της έκθεσης και οι τροπολογίες που θα υποβάλουμε θα είναι μικροβελτιώσεις, ουσιαστικά είναι επέστητες αλλαγές στην έκθεσή του. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τι επιπτώσει τη χρηματοπιστωτική κρίση ε, στο θέμα τη ισότητα των δύο φύλων, είπατε ήδη ότι η κρίση θα έχει περισσότερα μακροπρόθεσμες παρά βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να επιμείνουμε στο θέμα του δημοσίου χρέους ε, που θα πρέπει να τελεί στενό έλεγχο γιατί αν έχουμε χρέος, υπερχρέωση του δημόσιου φορέα και μεγάλο δημόσιο χρέος ε, θα πληγούν πάνω απ' όλα οι γυναίκες πιστεύω γιατί είναι αλληλένδετα τα δύο θέματα. Τώρα μακροπρόθεσμα η καλύτερη προστασία των γυναικών έναντι της φτώχειας και της ανεργίας είναι η κατάλληλη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και η σωστή αμοιβή τους, ε, αντίστοιχη με την αμοιβή των ανδρών για την ίδια εργασία. Όλα αυτά τα θέματα, όπως είπα, είναι αλληλένδετα και είπατε ότι χαιρόμαστε που νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι γυναίκες, αλλά αυτό είναι το απολύτως απαραίτητο, είναι το ελάχιστο. Πώς θα επιχειρηματολογούμε εμείς για πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και δίκαιη αμοιβή, αν δεχόμαστε η, η πολιτική ηγεσία της Ένωσης και οι θύνουσες θέσεις να μην στελεχώνονται ισότιμα από άνδρες και γυναίκες. Εμείς θα πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα για όλες τις νεαρές γυναίκες στην Ευρώπη και να δείξουμε ότι η συμμετοχή στην αγορά εργασίας είναι πολύ θετική και εξασφαλίζει και την οικονομική τους ανεξαρτησία. Και μακροπρόθεσμα αυτή είναι η καλύτερη προστασία κατά της κρίσης. Σε ό,τι αφορά το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, το επισήμανε ο εισηγητής μας και αυτό συζητήσαμε πριν από λίγο στην πολιτική μου ομάδα και πραγματικά άκουσα παραδείγματα χωρών όπου το μισθολογικό χάσμα όχι μόνο δεν γεφυρώθηκε, αλλά διευρύθηκε μέχρι και 40%. Εξοργιστικό και πολύ ανησυχητικό στοιχείο για πολλές χώρες. είναι απίστευτο. Αυτό καλό θα ήταν να το επισημάνουμε στην έκθεση. Άλλωστε, στο θέμα αυτό καλό θα ήταν να εγγύψουν και τα συνδικάτα, γιατί Μπορεί να έχουμε νομοθεσία για ίσα δικαιώματα, αλλά οι διαπραγματεύσει ε, για παρόμοιε αμοιβέ είναι στα χέρια των εργαζομένων και των εργοδοτών, των συνδικάτων και των εργοδοτών. Σε ό,τι αφορά την νομοθεσία που δεν συνιστά διακριτική μεταχείριση κατά των γυναικών, θα ήθελα να προσθέσουμε μία παράγραφο που να αναφέρεται στο γεγονός ότι Ακόμη και τώρα, ακόμη και στα νομοσχέδια που εξετάζει το, Συμβούλιο και, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, ισχύουν κάποιες εξαιρέσεις από την αρχή της μη διάκρισης. Και συνήθως αυτές οι εξαιρέσεις προβλέπονται για θρησκευτικούς λόγους. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε προσεκτικά, γιατί στην πατρίδα μου κάποια ε, θρησκευτικά σχολεία ή θρησκευτικά ιδρύματα είναι ελεύθερα να προβαίνουν σε διακριτική μεταχείριση κατά των γυναικών με το πρόσχημα της ε, ανεξιθρησκείας. Βέβαια η ανεξιθρησκεία είναι αναπαλωτρίωτο και θεμελιώδης ατομικό δικαίωμα που το προσπίζουμε, αλλά αυτό δεν δίνει δικαίωμα σε κάποια θρησκευτικά ιδρύματα ή θρησκευτικά σχολεία να προβαίνουν σε διακριτική μεταχείριση για αυτό το λόγο. Στη Γερμανία, ο, μεγαλύτερος, ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης είναι ο τομέας των σταθμών, παιδικών σταθμών, οι φροντίδες που κυρίως διαχειρίζονται εκκλησίες. Αυτό τους δίνει δικαίωμα να κάνουν διακρίσεις κατά των γυναικών. Αυτό να το προσέξουμε λοιπόν. Δεν θα πρέπει η θρησκεία να γίνεται λόγος για διάκριση. Επίσης, ό,τι αφορά τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, είναι πολύ ευαίσθητο αυτό το θέμα, αλλά αν δεν μπορούμε καν να αναγνωρίσουμε την αυτονομία των γυναικών στα θέματα αυτά, το δικαίωμα να αποφασίζουν για το σώμα τους, πώς είναι δυνατόν να καταπολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών, αν δεν τολμούμε καν να αναγνωρίσουμε την αυτονομία τους και το δικαίωμα να εξουσιάζουν το σώμα τους, Πώς ε, να πούμε όχι δεν θα τις χτυπάτε. Θα πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε την αυτονομία και τη σωματική ακαιρεότητα των γυναικών συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Τώρα, ευχαριστούμε κυρία Ιντβέλτ. Η επόμενη στον κατάλογο των ομιλητών είναι η κυρία Φιγκερέντο και μετά η κυρία Λούλινγκ. Πρώτα η κυρία Φιγκερέντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο εισηγητής μας ήδη στην έκθεσή του επέσε την προσοχή μας στις ε, συνέπειες που είχε η χρηματοπιστωτική κρίση στη ζωή των γυναικών. Εγώ θα ήθελα να αναπτύξουμε πιο διεξοδικά αυτό το θέμα και θα προτιμούσα η έκθεση να αντανακλά αυτές τις ανησυχίες μας. Γιατί η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή οι γυναίκες είναι αυτές που απολύονται, που απειλούνται με ενεργεία. Και σε μερικά εργοστάσια εργάζονται αμυστοί, γιατί υπάρχουν κάποιοι βιομηχανικοί κλάδοι που αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες και πολυεθνικές στην υποδηματοπία, στην κλωστοϊφαντουργία, στην βιομηχανία ένδυσης υπάρχουν προβλήματα και χιλιάδες γυναίκες ε, εργάζονται μισθή πάνω από χίλιες γυναίκες σε διαφορετικά εργοστάσια και επιχειρήσεις ε, στη χώρα μου μου είπαν την περασμένη εβδομάδα ότι δεν έχουν λάβει ακόμα τους μισθούς τους που ούτως ή άλλως είναι πενιχροί είναι γύρω στα 500 ευρώ το μήνα, αλλά ακόμη και αυτά τα 500 ευρώ ε, έχουν να τα, έχουν ε, λαμβάνουν από τον Οκτώβριο και βρισκόμαστε τέλη ε, Νοεμβρίου. Έχουν ούτω ή άλλω ελάχιστου μισθού και παρόλα αυτά ούτε αυτού δεν παίρνουν, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν τεράστια οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα. Και επιπλέον φοβούνται ότι θα κλείσουν και όλα αυτά τα εργοστάσια και επιχειρήσει και θα μείνουν στο δρόμο. Οι βιομηχανίες λοιπόν επηρεάστηκαν από την κρίση, έχουν πληγεί και μάλιστα τα θύματα αυτής της κατάστασης πρώτα απ' όλα είναι οι γυναίκες, οι εργαζόμενες της επιχειρήσης αυτές. Οι γυναίκες είναι αυτές που κατεξοχήν εργάζονται σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης ή σε σούπερ μάρκετ και μεγαλοκαταστήματα όπου οι γυναίκες εργάζονται είτε με μερική απασχόληση είτε εποχιακά είτε με συμβάσεις ε, ορισμένου χρόνου αλλά πολύ βραχυπρόθεσμες και εκεί οι γυναίκες απολύονται μαζικά χωρίς να έχουν καμία δυνατότητα ανέβρεσης θέσης εργασίας. Και αυτό επιδεινώνει όχι μόνο την κατάσταση στην απασχόληση αλλά και στο βιωτικό επίπεδο. Γιατί επειδή πολλές γυναίκες είχαν επισφαλή θέση απασχόληση δεν δικαιούνται καν επίδομα ανεργίας. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα σε ορισμένες χώρες. Εγώ σας μιλάω για καταστάσεις που γνωρίζω προσωπικά από την Πορτογαλία. Και όλα αυτά οφείλονται στην κρίση. Και δεν νομίζω ότι η Πορτογαλία είναι μια απομονωμένη περίπτωση. Σίγουρη και άλλες χώρες αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Γι' αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η εποχιακή, η μερική απασχόληση, η επισφαλής απασχόληση, η απασχόληση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου πολύ βραχυπρόθεσμες, είναι μορφές εργασίας που πλήττονται κατεξοχήν από την κρίση και τα πρώτα θύματα αυτής της κατάστασης είναι οι γυναίκες. Γιατί οι γυναίκες κυρίως εργάζονται σε κακοπληρωμένες ε, και ε, επισφαλείς θέσεις εργασίας. Θα πρέπει επίση να τονίσουμε την ανάγκη να συνδράμουμε επιχειρήσεις ή βιομηχανίες στις οποίες εργάζονται κυρίως γυναίκες ή να υποστηρίξουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν κυρίως γυναίκες στον τομέα των υπηρεσιών στον εμπορικό τομέα. Και όπως είπε και ο εισηγητή μα, να εξετάσουμε ιδιαίτερα το θέμα των ε, κρατικών υπηρεσιών, γιατί η συρρήκνωση του κρατικού προϋπολογισμού και οι περικοπές που γίνονται στον προϋπολογισμό ε, υπό το πρόσχημα της στήρησης ε, του Συμφώνου Σταθερότητας θα οδηγήσουν σε πολύ μεγάλη επιδείνωση κατάστασης, σε μια συγκυρία που είναι ήδη αρνητική. Και έτσι δεν θα επιδεινωθεί μόνο η κατάσταση των γυναικών που εργάζονται σε αυτούς τους κλάδους, αλλά θα επιδεινωθεί η παιδεία και θα χειροτερεύσει η κατάσταση σε πολύ σημαντικού κλάδου ε, κοινοφελής όπως είναι η υγεία, η παιδεία και που συμβάλλουν στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Όλα αυτά μας τα είπε ακροθυγός ο εισηγητής μας, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να τα αναπτύξουμε πιο διεξοδικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. κυρία Φιγκουρέντο. Και έτσι λοιπόν ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Λούλινγκ, η οποία είναι και η μόνη ευρωβουλευτής η οποία ε, είναι και παράλληλα και κοσμήτωρας. Κύριε Λούλινγκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω στον κύριο Ταραμπέλα ότι εξεπλάγει θετικά από την καλή ποιότητα της έκθεσής του. Έχουμε συνηθίσει σε αυτήν την Επιτροπή σε κάποιες εκθέσεις πολύ λιγότερο σωστά διαρθρωμένες από πλευράς κάποιων συναδέλφων ανδρών και γυναικών της πολιτικής του ομάδας. Παρ' όλα αυτά κάποιες παρατηρήσεις θα πρέπει να γίνουν και υπάρχουν και ορισμένα παράδοξα θα έλεγα τα οποία θα ήθελα να υπογραμμίσω. Να ξεκινήσω με μία παρατήρηση στα λεγόμενα της προλαλήσας σας. Αν υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρώνουν τις επιχειρήσεις, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Στρασβούργου. Αυτό είναι αρμοδιότητα του εργατικού δικαίου στις συγκεκριμένες χώρες. Είναι θέμα συλλογικών διαπραγματεύσεων και τώρα μην απαιτείται να ασχολούμεθα εμείς με κάθε επιχείρηση η οποία ίσως συλλογικων διαπραγματευσεων και τωρα μην απαιτειτε να πληρώσει τους εργαζομένους της. Έχουμε συγκεκριμένους κανόνες προς την κατεύθυνση αυτή και στα πλαίσια των συλλογικών διαπραγματεύσεων και στα πλαίσια του εργατικού δικαίου. Πέραν τούτου, να κάνω μία παρατήρηση σχετικά με την αιτιολογική σκέψη Β. Συμφωνώ να λέμε ότι Υπάρχουν περισσότερες γυναίκες που ασχολούνται με την επιμέρους απασχόληση και υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που το επιθυμούν αυτό. Ενθυμούμε ότι κάποτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδιαίτερα στη δική μου χώρα είχαμε διεκδικήσεις ακριβώς για να διεκδικήσουμε περισσότερες δυνατότητες επιμέρους απασχόλησης σε γυναίκες και σε άνδρες φυσικά που εθελοντικά θα ήθελαν να απασχοληθούν με τον τρόπο αυτό με τώρα με αυτά τα οποία λέγεται ότι οι γυναίκες είναι πλειοψηφία στις δημόσιες υπηρεσίε, όχι σε όλα τα κράτη-μέλη. Είναι αλήθεια όμως ότι στην εκπαίδευση ισχύει κάτι τέτοιο. Πάντως στη δική μου χώρα, στο δημόσιο τομέα, Η αλήθεια είναι ότι αν είναι κάποιος δημόσιος υπάλληλο, δεν έχει πλέον ανησυχία, είναι μόνιμη θέση απασχόλησης, έχει καλή σύνταξη, αμείβεται καλά. Και αν πω ότι οι γυναίκες στην εκπαίδευση και στην υγεία είναι πλειοψηφία, τότε θα υπήρχε κίνδυνος θα έλεγα να πω ότι κινδυνεύουν από ένδια, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, οι γυναίκες οι οποίες δουλεύουν στον δημόσιο τομέα δεν αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο κίνδυνο. Στην αιτιολογική σκέψη γάμα τώρα. Οι συνταξιούχοι γυναίκες και οι χείρες είναι αυτές οι οποίες προστατεύονται με τον καλύτερο τρόπο σε αυτή τη φάση σχετικά με τα εισοδήματά τους. Στο Β πάντα δεν θα έλεγα ότι δεν έχουν υπάρξει βελτιώσεις των συνθήκων απασχόλησης. Ίσως να μην έχουν υπάρξει επαρκείς βελτιώσεις. Σίγουρα. Αλλά θα ήταν άδικο να περιγράψουμε την κατάσταση λέγοντας ότι δεν έχουν υπάρξει βελτιώσεις. Όταν αναφερόμεθα και για τη διαφορά της αμοιβή, μιλάμε για το η διαφορά αμοιβή, γιατί μόνο οι μέση όροι έχουν κάποιο νόημα και δείχνουν ποιες είναι πραγματικά οι διαφορές. Θυμίζω ότι από το 1975 υπάρχει μια οδηγία η οποία έχει χρησιμεύσει πάρα πολύ στη δική μου χώρα για την διασφάλιση της ισότητας των αμοιβών. Συνεπώς, δεν θα πρέπει κανείς να είναι απόλυτα αρνητικός και διαρωτώ με αν πράγματι έχουμε ανάγκη από νέες νομοθετικές προτάσεις για την εφαρμογή πάντα της αρχής της ίσης αμοιβή. Εφαρμόζεται η οδηγία αυτή. Οι γυναίκες μπορούν να εκμεταλλευτούν από τα μέσα που δίδει στη διάθεσή τους, που θέτει στη διάθεσή τους η οδηγία αυτή και μια μεταρρύθμιση της συγκεκριμένης οδηγίας διαρωτώ με αν θα είναι καλύτερη από την σημερινή κατάσταση. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχουμε κάνει σε σχέση με την ισότητα των ευκαιριών διαρωτώ με αν θα πρέπει να υπάρξει μια αναθεώρηση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι ίσως να εφαρμοστούν οι οδηγίες αυτές με σωστότερο τρόπο στο τέταρτο εδόφιο. Λέτε ότι έχουν περισσότερους τίτλους, τα 100 τίτλους που εκδίδονται πανεπιστημιακούς, οι γυναίκες έχουν την πλειοψηφία. Πότε, πού, θέλω διευκρινήσεις. Στο L, αγγλικό, θα πρέπει να προσθέσετε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις δύο θέσεις κλειδιά, τις οποίες μόλις δώσαμε σε γυναίκες σε μία γυναίκα μάλλον και σε ένα άνδρα. Στο 5 αναφέρεστε στη δημοσιονομική λιτότητα. Εγώ θα προτιμούσα να αναφερθούμε και στη δική μου χώρα θα προτιμούσα μια δημοσιονομική εξυγίανση και όχι λιτότητα. Και στο σημείο 7 εκ νέου αναφέρεστε στη μέση διαφορά των αμοιβών. Θα πρέπει όχι μόνο να λέμε ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά υπάρχουν και διαφορές ανάμεσα στους διαφορούς οικονομικούς τομείς. Στο σημείο 9. Λέτε και πολύ σωστά ότι απαιτείται μια καλύτερη μεταφορά των κοινοτικών ρυθμίσεων. Γιατί τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει τη δουλειά της. Γιατί αν πρέπει να ζητάμε κάθε φορά στα κράτη-μέλη να μεταφέρουν τις οδηγίες το ταχύτερο δυνατόν που αφορούν την ισότητα ανδρών και γυναικών ενώ οι οδηγίες αυτές είναι σε ισχύ από το 1975 αυτό δεν έχει νόημα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τη δουλειά της πραγματικά έτσι ώστε οι οδηγίες αυτές να εφαρμοστούν και να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη οι χώρες οι οποίες δεν έχουν εφαρμόσει σωστά στο εθνικό τους δίκαιο της διατάξης των οδηγιών. Δεν μου αρέσει λοιπόν αυτή η ιδέα δημιουργίας ε, ενός, μιας χάρτας ευρωπαϊκής για τα δικαιώματα της γυναίκας. Έχουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα μια χάρτα, καλύπτει και τις γυναίκες. Εσείς είσαστε κατά των διακρίσεων και τώρα θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή αυτή η ιδέα. Είναι μία από τις χειρότερες ιδέες τις οποίες είχατε στην μακρά σας πολιτική σταδιοδρομία. Για το 11. Να σας θυμίσω, έχοντας διαβάσει προσεκτικά το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά τις επαγγελματικές και τομεακές διακρίσεις, να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεχάσει ότι στη δεκαετία του 80, ήδη από τη δεκαετία του 80, είχε δημιουργηθεί ένα δίκτυο, ένα δίκτυο το οποίο, του οποίου ηγείτο τότε η κυρία Σιρό, πολύ γνωστή στη Γαλλία. Ήμουν εμπειρογνώμων στα πλαίσια αυτού του δικτύου στη δεκαετία του 80 ονομαζόταν πολλαπλασιασμός των επαγγελματικών επιλογών των νέων και των γυναικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρω τι συνέχεια έδωσε στην εργασία αυτή η οποία είχε κοστίσει αρκετά και το θυμάμαι πολύ καλά διότι και εγώ είχα ωφεληθεί από αυτό. Δεν σημαίνει βέβαια ότι η δική μου χώρα είναι μικρή και δεν αποφελείται. Λοιπόν, να ρωτήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτές τις εργασίες τι τις κάνει εν πάση περιπτώσει. Έχουν περάσει 30 χρόνια. Είχαμε κάνει τεράστιες εκθέσεις και για το Λουξεμβούργο. Μιλάμε χιλιάδες σελίδες. Τις έχω κάπου κρυμμένες στο σπίτι. Γιατί δεν δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέχεια. Η ίδια παρατήρηση ισχύει επίσης και για τη φτώχεια των γυναικών ιδιαίτερα όταν φτάνω στη στιγμή της συνταξιοδότησης. Οι συντάξεις απειλούνται, έχετε δίκιο και έχει δίκιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το υπογραμμίζει γιατί οι γυναίκες δούλεψαν λιγότερο σε μια στιγμή της ζωής τους γιατί έπρεπε να μείνουν λίγο στο σπίτι και επέλεξαν να μείνουν λίγο στο σπίτι για να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους και τιμωρούνται γι' αυτό σε επίπεδο συνταξιοδοτικό και αν θυμάμαι καλά το 85, το 95 συγγνώμη, μετά από δική μου πρωτοβουλία υπήρξε μια έκθεση η οποία έλεγε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια οδηγία για το λεγόμενο split των δικαιωμάτων των συνταξιδιωτικών σε περίπτωση ε, στάσης ε, εργασίας των γυναικών. Και στην Γερμανία αυτό είχε προχωρήσει ε, και ίσως δεν προχώρησαν οι άλλες χώρες, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ζήτησε την εφαρμογή αυτής της ρύθμισης. Καμία συνέχεια δεν δόθηκε. Γιατί κάτι τέτοιο θα επέτρεπε στις γυναίκες και στους άνδρες βέβαια. Υπάρχουν περισσότεροι άνδρες ε, τα τελευταία χρόνια που ασχολούνται με τα οικιακά και εγκαταλείπουν την επαγγελματική του δραστηριότητα, αλλά ο αριθμός δεν είναι ικανός ακόμη. Και αυτό δεν θα πρέπει να δημιουργεί προβλήματα τη στιγμή της συνταξιοδότησης. Δεν έχει δώσει, επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καμία συνέχεια στα ψηφίσματά μας αυτά. Και μετά ε, χύνει κροκοδίλια δάκρυα για την κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να τα θυμίσουμε όλα αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα επίσης να κάνω μία επιπλέον παρατήρηση. Ευτυχώς τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας προσκαλεί και ζητά ιδιαίτερα από τους νομοθέτες να επιταχύνουν τις διαδικασίες για τις προτάσεις που τροποποιούν την οδηγία για την γονική άδεια και για τους ανεξάρτητους και τις ανεξάρτητες μάλλον εργαζόμενες. Εμείς αυτό το είχαμε προχωρήσει, ξέρετε, εδώ και οκτώ μήνες. αλλά ούτε η Τσεχική Προεδρία ούτε η Σουηδική Προεδρία δεν ασχολήθηκαν σοβαρά με αυτό. Εμείς είχαμε ζητήσει στα πλαίσια της κοινή θέση να εφαρμοστούν αυτά που ζητάει η έκθεση από το μήνα Μάιο. Και η προστασία της μητρότητας είναι ένα σημαντικό θέμα και λόγω ακριβώς της ποιότητας της έκθεσης της κυρίας Εστρέλα με τις 73 τροπολογίες οι οποίες δεν βελτιώνουν το κείμενό της κάνουν απλά διακρίσεις ανάμεσα στη γονική άδεια, την πατρική άδεια, τη μητρική άδεια κτλ. Έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση και δεν καταλαβαίνω πώς θα καταλήξουμε σε μια αποδεικτή λύση, αποδεικτή και για το Συμβούλιο και διαπραγματεύσιμη με το Συμβούλιο εφόσον υιοθετήσουμε για μια ακόμη φορά μια τόσο χαοτική έκθεση, τόσο χαοτική όσο η τελευταία την οποία αναβάλαμε τη συζήτησή της και θα επανέλθουμε αύριο. Αυτές είναι οι λίγες παρατηρήσεις τις οποίες είχα να κάνω. Μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίες, αλλά πρέπει να τονίσω ότι η ποιότητα είναι καλή. Και θα πρέπει όμως να υπάρχουν κάποιοι παλαιοί σαν και μένα που υπενθυμίζουν ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχολούμεθα με θέματα τα οποία μόλις φαίνεται να ανακαλύπτει στην έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ για τα ίδια θέματα έχει ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για να δημιουργήσει δίκτυα, συμβούλους, εκθέσεις όλα αυτά έχουν γίνει, έχουν γίνει καλά νομίζω, αλλά δεν φαίνεται ίχνος τους κανένα σήμερα. Και θα πρέπει για να δούμε πραγματικά τις ανάγκες σε επίπεδο τοπικό και σε επίπεδο περιφερειακό και εθνικό να δούμε τι γίνεται με την φύλαξη των παιδιών σαν παράδειγμα που είναι ένα ε, θέμα σε εκκρεμότητα. Δεν ξέρω τι χρήματα έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να τα κατανείμουμε όπως θα έπρεπε. Δεν ισχύει συνήθως κάτι τέτοιο. Τα χρήματα τα οποία έχουν οι δήμοι και οι κοινότητες δεν είναι τόσο ψηλά όσο στο παρελθόν και δεν ξέρω τι πράγματι μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Αύριο λοιπόν θα επανέλθουμε σε αυτήν την έκθεση της κυρίας Εστρέλα και νομίζω ε, θα μπορέσουμε να ενημερωθούμε καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ για τις παρατηρήσεις. Η κυρία Έρνστ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως εδώ πρόκειται για ένα θέμα με πολλές κοινωνικές προεκτάσεις ε, και χαίρομαι πάρα πολύ που ο εισηγητής ε, προσπάθησε το θέμα αυτό να το συρρυκνώσει σε 21 σημεία. Βεβαίως ε, μπορώ να πιστέψω, θεωρώ ότι ήδη τώρα ότι δεν θα παραμείνει στα 21 σημεία, θα επεκταθεί η έκθεση. Δεν πειράζει, δεν είναι τόσο τραγικό. Σε αντίθεση με την προαλήσα, εγώ πρέπει να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που θα υπάρξει μια νέα νομοθετική πρόταση της Επιτροπής και για το πολύ ενδιαφέρον θέμα που είναι ίση αμοιβή για άνδρες και γυναίκες. Ομιλώ κάτω από το γερμανικό πρίσμα. Εμείς έχουμε μια χώρα όπου περίπου όπου έχουμε τις γυναίκες που για την ίδια εργασία πληρώνονται κατά 1 τέταρτον μέχρι και 1 τέταρτον λιγότερο από ότι οι άνδρες. Έτσι λοιπόν Υπάρχουν οι κανονισμοί, τους οποίους όμως κανείς δεν λαμβάνει υπόψη του για να το πω έτσι απλά. Άρα δηλαδή πρέπει να θεσπιστούν δεσμευτικές διατάξεις και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να καταφύγουμε στα δικαστήρια, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο των κυρώσεων. Θα το έβρισκα λοιπόν σωστό ε, να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης ε, χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι αναφέρεται ε, το θέμα της Ευρωπαϊκής Χάρτας δικαιωμάτων γυναικών. Βεβαίως ε, είναι σαφές ότι η Γαλλική Επανάσταση δεν έφτασε μέχρι τις γυναίκες. Οι γυναίκες αργότερα προστέθηκαν στις εξελίξεις, αργότερα θεωρήθηκε ότι και οι γυναίκες ε, είναι άνθρωποι. Θεωρώ λοιπόν ότι μια τέτοια χάρτα θα μπορέσει να δείξει το τι ακριβώς αφορά τις γυναίκες και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οι γυναίκες ε, στην ιστορία ε, ήταν πάντα ένα τμήμα κάποιου άλλου πράγματος. Τμήμα της οικογένειας, ε, μητέρα, τμήμα του παιδιού. Όμως ως γυναίκα η γυναίκα δεν βρίσκεται ποτέ ως ένα ανθρώπινο και είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να προσθέσω το εξή: Η συνάδελφός μου το ανέφερε ήδη. Θα πρέπει να αναφερθούμε ταχύτατα στο ότι η γυναίκες ε, δεν αμείβονται ικανοποιητικά. Στη Γερμανία έχουμε θέσεις εργασίας με πολύ κακές αμοιβέ που στο μεγαλύτερο βαθμό καλύπτονται από τις γυναίκες. Χωρίς κοινωνική ασφάλιση Πρόκειται λοιπόν για ένα τεράστιο πρόβλημα γιατί σε εμά δεν προβλέπεται και κατώτατος μισθός. Μιλάμε λοιπόν για πάρα πολλές γυναίκες με πολύ κακές αμοιβέ και το θέμα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω γυναίκες στις ηγετικές θέσεις. Εκεί πρέπει να είμαστε πιο σαφείς. Τι ακριβώς επιθυμούμε. Εγώ ε, προσωπικά ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε όσον αφορά τις ποσοστώσεις. Αλλιώς δεν θα οδηγηθούμε πουθενά. Το βλέπω λοιπόν στη Γερμανία. Έχουμε πολλές γυναίκες που έχουν πολύ καλύτερα πτυχία από τους ε, άντρες αλλά παρόλα αυτά δεν καταλαμβάνουν τις θέσεις που τους αξίζουν. Και μόνο το 10% των ε, καθηγητών είναι γυναίκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες είναι πιο χαζές, θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι καθηγήτριες. Υπάρχουν λοιπόν θέματα που πρέπει να τα εξετάσουμε. Και κατόπιν υπάρχουν και κάποια άλλα που λείπουν. Θα ήθελα δηλαδή εγώ να συμπεριλάβουμε μία παράγραφο για την κατάργηση αυτού του ε, πατριαρχικού μοντέλου ζωής. Υπάρχει, υπάρχει αυτό στο μυαλό μας ε, αυτή η ανισότητα ανδρών και γυναικών. Αυτή λοιπόν, αυτό το πατριαρχικό μοντέλο έχει επηρεάσει και την παιδεία. Πρέπει να δούμε λιγάκι το θέμα της παιδείας και κατά την άποψή μου ε, να ε, εξετάσουμε, να ε, κάνουμε μια πρόταση οι γυναίκες και οι άνδρες να βρίσκονται στην ίδια μοίρα ε, και αυτά να μην είναι απλά ένα όνειρο θερινής νυχτός. Τέλος, τελευταίο σημείο, γυναίκες με αναπηρία. Γνωρίζω από τη δουλειά μου στον τομέα αυτό ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες που έχουν αυτή την ε, διπλή δυσάρεστη θέση. Πρέπει να δούμε λοιπόν αν μπορούμε να κάνουμε κάτι έτσι ώστε η θέση αυτών των ε, γυναικών ε, που έχει σχέση και με την εργασία αλλά και με άλλε συμπεριφορές διακριτική μεταχείρισης να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προσθέσουμε κάποια θέματα στην έκθεσή μα. Η ε, προλαλήσα αναφέρθηκε και στο θέμα γυναίκα και σύνταξη. Σωστά. Και αυτό πρέπει να το δούμε πιο συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι ότι η ανατροφή των παιδιών είναι κάτι που θα πρέπει να συνυπολογίζεται στη σύνταξη. Αυτό λοιπόν πρέπει να το γράψουμε. Δεν είναι αυτονόητο, θεωρώ ότι ε, αυτό βέβαια έχει άμεση σχέση και με τον πλούτο και την φτώχεια. Ε, τελειώντας θα ήθελα να πω ότι εμείς ε, προτιθέμεθα να καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες και νομίζω ότι η συζήτηση μέχρι τώρα διεξήχθη περισσότερο από ικανοποιητικά. Σας ευχαριστούμε κύριε Άρνστ. Όντω βρισκόμαστε μέσω μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ε, θα δώσω το λόγο στην κυρία Κορνέλισεν και μετά στην κύριο Σιμάνσκι. Ευχαριστώ. Όπω και οι προλαλήσεις θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον ε, εισηγητή μα γιατί η έκθεση του πραγματικά είναι πολύ μεστή και περιεκτική. Θα υποβάλουμε βέβαια κάποιες τροπολογίες, αλλά ουσιαστικά είναι μικρές προσθήκες στην ε, έκθεσή του. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο τεινά. Στην έκθεση αναφέρεται καλύτερη εφαρμογή των υπαρχουσών καταθετηρίων γραμμών και πολιτικών. Αυτό νομίζω ότι έχει κεφαλαιόδη σημασία και θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Γιατί η ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα για τις γυναίκες και απτές συνέπειες μόνο εφόσον εφαρμοστούν θα πρέπει να στυλιτεύσουμε τα κρατη να κατονομάσουμε όσους δεν εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία, να επιβραβεύσουμε αυτούς που το κάνουν. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Τα θέματα της ε, συμμόρφωσης και της σωστής εφαρμογής. Αναφέρεται ε, το θέμα της κρίσης και της αλλαγής στην αγορά εργασίας. Η κρίση μπορεί να δώσει και κάποιες ευκαιρίες, προς το παρόν όμως δημιουργεί και πολλές απειλές στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και είναι πολύ θετικό ε, που αναφέρουμε τις συνέπειες που θα, έχω, θα έχει στην κατάσταση των γυναικών ε, η συρρήκνωση του εθνικού προϋπολογισμού και θα πρέπει οι περικοπές που θα γίνουν στους κρατικούς προϋπολογισμούς να μην επικεντρωθούν στις ε, δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικές, κάτι που θα πλήξει ακόμη περισσότερο τη θέση των γυναικών. Λαμβάνονται κάποια μέτρα για να αμβληθούν οι συνέπειες της κρίσης και να δοθούν κίνητρα εξόδου από αυτήν. Έχω πάντως την υπόνοια ότι δυστυχώς πολλά αυτά τα κονδύλια θα φτάσουν σε ανδρικά χέρια στους ανδροκρατούμενους τομείς και δυστυχώς δεν θα ωφελήσουν τις γυναίκες που και αυτές πλήττονται άμεσα από την κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια σωστή κατανομή μεταξύ των δύο φύλων στα κονδύλια για την καταπολέμηση της κρίσης και την οικονομική ανάκαμψη. Θα πρέπει επίσης ε, να βοηθήσουμε τις γυναίκες να παραμείνουν στην αγορά εργασία. Έχουμε όμως και το πρόβλημα της γύρεσης του πληθυσμού. Βέβαια, αυτό το πρόβλημα είναι κάπως πιο μακροπρόθεσμο. Είναι μια πιο μακροπρόθεσμη κοινωνική αλλαγή που θα επηρεάσει και τις γυναίκες με διαφορετικό όμως τρόπο από ό,τι τους άντρες. Και σίγουρα θα χρειαστούμε και άνδρες και γυναίκες στην αγορά εργασίας για να καλύψουν τις κοινέ θέσεις που θα απομείνουν από τη γύρανση του πληθυσμού. Και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε και συμπληρωματικά μέτρα, ώστε να γίνουν οι μισθοί πιο ελκυστικοί για τις γυναίκες, να υπάρξουν μέτρα για τις άδειες πατρότητας και μητρότητας, φύλαξης και φροντίδας των παιδιών, πιο ελαστικό ωράριο εργασίας και μέτρα για καλύτερη, καλύτερο συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ε, ζωής, ώστε να αισθάνονται άνετα στην αγορά εργασίας και άνδρες και γυναίκες και να παραμείνουν όσο το δυνατό περισσότερο γίνεται. Ίσως θα πρέπει να συντάξουμε και δική παράγραφο για τις συνέπειες της γύρας του πληθυσμού, ειδικά στις γυναίκες. Επίσης, θα πρέπει να εφαρμόσουμε εμπράκτος τη στρατηγική της Λισαβόνας. Βέβαια αυτός είναι πιο μακροπρόθεσμος ε, στόχος και θα πρέπει σίγουρα να ε, συμπληρωθεί και με ένα κεφάλαιο ισότητας. Αυτά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κορνέλησεν. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Σιμάνσκι και μετά η κυρία Τόμσον. Ο κύριος Σιμάνσκι. Χωρίς μικρόφωνο. Πρέπει να τα επαναλάβω μάλιστα γιατί δεν ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο. Θα ήθελα και εγώ να επικροτήσω την έκθεση του κυρίου Ταραμπέλα και ε, πιστεύω ότι θα πρέπει σε αυτό τον ευρύ αγώνα για τα δικαιώματα της γυναίκας να επικεντρωθούμε σε ορισμένα θέματα που δεν είναι επίμαχα και αφιλεγόμενα, είναι προφανή και παρόλα αυτά δυστυχώς εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται και αυτό είναι πολύ σκαδαλώδες και εξοριστικό. Για παράδειγμα, έχουμε γυναίκες που είτε από επιλογή είτε από αναγκαιότητα ένα μεγάλο τμήμα της ζωής τους ε, και της ενέργειάς τους την αφιερώνουν στην ανατροφή των παιδιών. Βέβαια εδώ ε, αναφέρθηκε κάποια κριτική προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να περάσει από τα λόγια στα έργα και να κάνει μια επισκόπηση της νομοθεσίας των κρατών μελών προτείνοντας ε, κάποιες ε, ελάχιστες διατάξεις προστασίας αυτών των γυναικών, γιατί η κατάσταση σε ορισμένες χώρες είναι τραγική και πραγματικά αυτό είναι σκανδαλώδες. Δεύτερον, σίγουρα υπάρχει μεγάλη ανώμια μορφία μεταξύ της συζήτησης, των γνωμοδοτήσεων, των διασκέψεων, αυτών που θεωρητικά συζητούμε σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει με... μεγάλη διαφορά λοιπόν μεταξύ αυτής της θεωρίας αλλά και της πράξης, γιατί στην πράξη οι γυναίκες ε, υφίστανται διακριτικές μεταχειρήσεις ε, και αρνητική διάκριση. Ακόμη και στις ηγετικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμμετοχή των γυναικών είναι ελάχιστη. Και αυτό είναι φανές ότι υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ των ε, αγαθών προθέσεων και των, των βαρύγδουπων δηλώσεων και της πρακτικής εφαρμογής τους. Και μπορεί αυτή η άποψη να μην και πολύ δημοφιλής, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι φιλόδοξες και ε, ικανές γυναίκες έχουν δικαίωμα να καλύψουν κάποιες ηθήνουσες και ηγετικές ε, θέσεις. Παρόλα αυτά δεν έχουν τέτοια δυνατότητα. Ακόμη και στα κοινοτικά θεσμικά όργανα υπάρχει διάκριση κατά των γυναικών και μικρή συμμετοχή του, ιδιαίτερα σε ηθήνουσε και ηγετικέ θέσει. Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασία. θα ήθελα να πω ότι πολλέ γυναίκε σε πολλέ χώρε ε, αναλαμβάνουν κάποιες θέσεις, ε, όχι μόνο ε, ανάλογα με τις ικανότητές τους, τις γνώσεις, τις δεξιότητές τους και την αυτοεκπλήρωσή τους, αλλά και για οικονομικούς λόγους. Γιατί αν κάποιος θέλει μία δουλειά ανάλογα με τη μόρφωσή του, έχει δυνατότητα επιλογής, δεν εξαναγκάζεται να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά πολλές γυναίκες σε φτωχότερε χώρες με δινή οικονομική κατάσταση δεν έχουν δυνατότητα επιλογής. Ε, ό,τι δουλειά βρουν θα τη δεχτούν και αυτές είναι δυστυχώς θέσεις ε, κακοπληρωμένες αλλά από ανάγκη οι γυναίκες ε, τις δέχονται. Ε, θα ήθελα να εκφράσω την επιθυμία αυτή η έκθεση να μην παραμείνει στα χαρτιά, αλλά πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια επισκόπηση τη κοινοτική νομοθεσία και των κρατικών νομοθεσιών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το θέμα το συνταξιοδοτικό για τι γυναίκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Τόμψον, πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή για τη δουλειά του και νομίζω ότι πραγματικά μας καταθέσετε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Ε, βασικά θέματα κομβικής σημασία που αφορούν στην ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Εγώ έχω μόνο λίγα σχόλια να κάνω. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι αυτά που είπε ο κύριος Φιγκερέντο, η κυρία Φιγκερέντο για την κρίση με εντυπωσίασαν. Ε, η κρίση πλήττει επιφανειακά και τους άνδρες και τις γυναίκες. Ε, ε, σε, στο δικό μου, στη δική μου την πατρίδα στον οικοδομικό τομέα απολύθηκαν και πάρα πολλοί άντρες. Βεβαίως, όσο βαθαίνει η κρίση, μειώνονται και οι δημόσιες δαπάνες και αυτό ε, αφορά τις ε, γυναίκες ως εργαζόμενες στο δημόσιο τομέα, αλλά και ως ε, αποδέκτες υπηρεσιών από το δημόσιο τομέα αποδέκτριε μάλλον. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε παραδείγματα της βαριά ε, βιομηχανία που υπέστη τεράστιο πλήγμα και εκεί ε, το πλήγμα ήταν κυρίω για τους άνδρες. Σε χώρες όμως όπου υπάρχει ε, βαριά βιομηχανία, όπως είπε η κυρία Φιγκερέντο, στην Πορτογαλία δεν υπάρχει βαριά βιομηχανία και η ελαφριά βιομηχανία που βλέπουμε σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ε, στα νέα. Η ε, ελαφριά αυτή βιομηχανία αφορά κυρίως τις γυναίκες. Αυτές εργάζονται εκεί και αυτές ε, πλήττονται από την κρίση. Όταν λοιπόν συζητάμε το θέμα κατά πόσον επηρεάζονται περισσότερο οι άνδρες ή οι γυναίκες από την κρίση, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε κατά νου και την διαφορετικότητα των καταστάσεων. Αυτά όλα είναι συνάρτηση του για ποιο κράτος μέλος μιλάμε. Είναι δύσκολο λοιπόν να γενικεύσει κανείς και να αποφανθεί γενικά για την Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα τη διαφορά στην αμοιβή ανάμεσα στα δύο φύλλα. Η διαφορά αυτή αντιμετωπίζεται από τους κοινωνικούς εταίρους στην Ευρώπη. Όμως πρέπει να έχουμε κατά νου, και νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό, στην σχετική οδηγία η ευθύνη δεν βρίσκεται στα χέρια των ε, κοινωνικών εκτέρων. Δεν είναι αυτοί οι αρμόδιοι για να μειώσουν αυτή τη διαφορά αμοιβή. Η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη. Εκείνη καλείται να εξηγήσει, να εκπαιδεύσει, να διασφαλίσει ότι πράγματι μειώνεται το χάσμα των αμοιβών μέσα από τις ε, συλλογικές διαπραγματεύσεις. Και αυτό έχει σχέση και με την εφαρμογή της οδηγίας. Με το κατά πόσο δηλαδή μια κυβέρνηση εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στον τομέα αυτό. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε κυρία Τόμσον. Η κυρία Ουβή έχει το λόγο. Θα ήθελα κι εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα έκθεσή του. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, κυρίως ε, γιατί ε, συντάχθηκε από έναν άντρα. Στην Εστονία κάτι τέτοιο τουλάχιστον με, τώρα θα ήταν αδύνατον. Να αναφερθώ σε κάτι, αν μου επιτρέπετε, που θέλω εκεί να υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες. Γνωρίζουμε ότι στην Ευρώπη σιγά σιγά έχει αλλάξει το πρότυπο της οικογένειας οι ε, μονογονικές οικογένειες δεν είναι πια κάτι το ιδιαίτερο και ούτε και ενοχλούν και κανένα. Όμως ε, οι πατέρες ε, σε πολλά κράτη-μέλη εξακολουθούν να μην εκπληρούν τις υποχρεώσεις τους. Οι μητέρες δεν στηρίζονται από τους πατέρες για να αναθρέψουν τα παιδιά τους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό επειδή σήμερα διατρέχουμε αυτή την κρίση, το θέμα αυτό να αναφερθεί περισσότερο στην έκθεση. Παραδείγματο χάρη θα μπορούσε να προταθεί το κράτος να αναλάβει προσωρινά το καθήκον στήριξης ε, της μητέρας αν δεν το κάνει ο πατέρας. Και το κράτος αργότερα μπορεί να διεκδικήσει χρήματα από τον πατέρα για αυτή του την προσφορά. Ε, κάτι άλλο που ενδιαφέρει είναι ε, γυναίκες με αναπηρία. Οι γυναίκες αυτές ποτέ δεν εκπροσωπήθηκαν ικανοποιητικά στην αγορά εργασίας. Κυρίως σήμερα η διαφορά αυτή, το χάσμα που υπάρχει, επιτείνεται. Σε γενικές λοιπόν γραμμές θα έλεγα ότι μου αρέσει πάρα πολύ η έκθεση, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια σημεία όπου πράγματι θα μπορούσαμε να προβούμε σε κάποιες ε, βελτιώσεις. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αβή. Δεδομένου υπάρχει πρόσωπο Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ήθελε να λάβει το λόγο. Όχι. Καλώ. Τότε θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή μα, τον κύριο Ταραμπέλα, για τα σχόλιά του μετά αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε για την έκθεσή του. Σας ευχαριστώ. Δεν πρόκειται να επαναλάβω όλες τις παρατηρήσεις. Φυσικά αυτό που με ικανοποίησε ήταν η ιδιαίτερη εκτίμηση που, έδωσαν, που έδειξαν οι συνάδελφοι που επισήμαναν ε, την ισορροπία που έχει έκθεσή μου και μάλιστα μοιράστηκα αυτή τη χαρά με την, ε, ε την Κριστίν Ραμό, την ε, συνεργάτη μου που πριν από λίγο καιρό είχε γράψει και ένα βιβλίο για τις γυναίκες και δεν περίμενα να την κατανομάσω, αλλά θα ήθελα να την επενέσω και μοιράστηκα μαζί της αυτή τη χαρά. Μιλήσαμε για το ότι η κοινοτικοί φορείς θα πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα και δεν θα πρέπει εμείς να κοκκινίζουμε από ντροπή, ε, γιατί θα πρέπει στο, δημόσιο γυναίκες και στη, στα κοινοτικά όργανα να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή και να μην υπάρχουν μισθολογικές διαφορές. Βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε τέτοιες διαφορές μισθολογικές. Περισσότερο στον ιδιωτικό κλάδο υπάρχουν διαφορές, γιατί μεγάλες επιχειρήσεις εφαρμόζουν ε, μισθολογική διάκριση κατά των γυναικών. Και επίσης υπάρχει πολύ μικρή συμμετοχή γυναικών σε διευθυντικές θέσεις, αλλά περισσότερο αυτό συμβαίνει στον ιδιωτικό κλάδο, στο δημόσιο, ούτε στα κράτη-μέλη υπάρχουν τέτοιε μισθολογικέ διαφορέ. Η κυρία Φιαγκερέντο και η κυρία Τόμσεν ε, μίλησαν για τις επιπτώσεις που είχε η κρίση ε, στις διάφορες χώρες. Ε, στη βαριά βιομηχανία θύματα περισσότερο είναι οι άνδρες, ενώ στην ελαφριά οι γυναίκες. Αλλά και όταν γίνεται αναδιάρθρωση των κοινωνικών κοινοφελών υπηρεσιών, εκεί πλούνται ιδιαίτερα οι γυναίκες. Ε, φυσικά υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών και αυτό θα πρέπει να το επισημάνουμε. Η κυρία Λούλινγκ επισήμανε ε, το γεγονό ότι η έκθεση μου είναι αρκετά εύστοχη και χαίρομαι ιδιαίτερο. Βέβαια, από αυτά που είπε προέκυψαν κάποιες ε, αντιφάσεις, αλλά για το θέμα της μερική απασχόλησης, για παράδειγμα. Όντως, όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν τη μερική απασχόληση, αλλά μερικές φορές το κάνουν από ανάγκη και όχι από ελεύθερη επιλογή. Και μάλιστα, σε ένα νοικοκυριό με τους δύο γονείς που εργάζονται και οι δύο, όταν, κάποιο, όταν γεννιέται ένα παιδί, αν έχει αναπηρία ένα παιδί, θα πρέπει οι γονεί να διαλέξουν ποιο από του δύο θα θυσιαστεί και θα περνάει περισσότερε ώρε στο σπίτι για να φροντίσει τα παιδιά, να αναθρέψει τα παιδιά, όταν υπάρχει και σοβαρή αναπηρία. Συνήθως είναι η γυναίκα αυτή που αναγκάζεται να μείνει στο σπίτι και να ασχοληθεί με τα παιδιά και να διακόψει την επαγγελματική της σταδιοδρομία, ενώ ο σύζυγος ε, την ε, συνεχίζει τέτοιες ευθύνε, κυρίως οικογενειακές, αναλαμβάνουν περισσότερο οι γυναίκες. Σε ό,τι αφορά τις ε, πολυάριθμες παρατηρήσεις κυρίας Λούλινγκ, αλλά και άλλων συναδέλφων, θα ήθελα να πω ότι ε, μην ξεχνάτε την προθεσμία για τις τροπολογίες που λύγει την επόμενη Δευτέρα και θα δεχτώ τις τροπολογίες που θα διευκρινίσουν καλύτερα κάποια σημεία της έκθεσης. Ό,τι αφορά τις μισθολογικές διαφορές, η κυρία Ένς επισήμανε αυτό το θέμα, το 25% που ισχύει στη Γερμανία. Ε, όταν αναφέρω το 17% δεν έλαβε υπόψη την μερική απασχόληση, που μερικές φορές είναι μία ανάγκη για τις γυναίκες και όχι ελεύθερη επιλογή. Και στην, στο δημόσιο τομέα, όπως είπε η κυρία Ιντβέλτ, είναι αλήθεια ότι στο δημόσιο τομέα υπάρχουν διαφορές, αλλά πολύ χειρότερες διαφορές υπάρχουν στις ε, επιχειρήσεις πολυεθνικές, ε, που ελάχιστες γυναίκες έχουμε σε διευθυντικές θέσεις, ενώ στο δημόσιο τομέα είναι γύρω στο 10%. Αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να επιφέρουμε κάποιες μεταρρυθμίσεις. Για το πατριαρχικό σύστημα, αυτά είναι τα στερεότυπα που ισχύουν, που μερικές φορές είναι αμφίδρομα, Ίσως θα πρέπει να, ενημερώσουμε, να οργανώσουμε και ενημερωτικέ εκστρατείε για να αφυπνίσουμε τους νέους στα σχολεία, γιατί εκεί είναι που γεννιόνται τα στερεότυπα και προκαταλήψεις από τα σχολικά εγχειρίδια. Από εκεί θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε την αλλαγή της νοοτροπίας. Από τη σωστή διαπαιδαγώγηση ήδη από τη σχολική ηλικία. Η καλύτερη εφαρμογή των ε, εφισταμένων πολιτικών είναι απαραίτητη πριν προβούμε σε μεταρρυθμίσεις. Αντί να υποβάλουμε νέες προτάσεις, καλύτερα να εφαρμόζουμε σωστά τα υπάρχοντα κείμενα. Σωστά και μάλιστα πέρσι είχα ε, ασχοληθεί με τη μεταφορά μιας οδηγίας ε, που πέρασε έξι αναγνώσεις στην κυβέρνηση Βαλονίας, γιατί στο μεταξύ υιοθετήθηκαν και νέε κοινοτικέ οδηγίες και μέχρι να περάσει από τη διαδικασία την κοινοβουλευτική και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση χρειάστηκε να περάσει από έξι διαδοχικέ αναγνώσει γιατί στο μεταξύ είχε αναθεωρηθεί. Καλύτερα λοιπόν έχουμε λιγότερη νομοθεσία καλύτερη νομοθεσία και φυσικά καλύτερη και σωστότερη εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας. Κύριε Σιμάνσκι, ευχαριστώ για τα συγχαρητήριά σας. και όταν μίλησε για γυναίκες που επιλέγουν να παραμείνουν στο σπίτι, μίλησε όμως για ταλαντούχες και ικανές γυναίκες. Ίσως ε, τη στιγμή που ε, θα ε, θα διοριστεί μία ανίκανη γυναίκα σε μία ηθήνουσα θέση, τότε είναι που θα, θα, δεν θα έχει πια λόγο ύπαρξη αυτή η επιτροπή. Γιατί όντω <laughs> ανίκανοι άνθρωποι πολλέ φορέ ορίζονται σε τέτοιε θέσει. Δεν ξέρω τα private joke αυτό, κύριε Σιμάνσκι. Κύριε Τόμσεν, σας ευχαριστώ για το επένους. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ βαριάς και ελαφριάς τροποθεσίας και ποια είναι τα θύματα της κρίσης στην κάθε περίπτωση. Πάντως υπάρχουν διαφορές και μεταξύ των διαφόρων περιοχών και μεταξύ των διαφόρων χωρών και μεταξύ των διαφόρων κλάδων της βιομηχανίας. Γι' αυτό και θα πρέπει η ανάλυση που θα κάνουμε να είναι πιο σαφής. Τώρα για τι ε, ανήπαντρε γυναίκε ή τι μονογονεϊκέ οικογένειε, αυτό πια σήμερα είναι συνηθισμένο φαινόμενο, ενώ πριν από μερικά χρόνια ήταν η εξαίρεση και δημιουργούσε αμηχανία. Αλλά έχουμε και το θέμα των πατέρων που αποποιούνται των ευθυνών του, γιατί μένουν οι γυναίκε πολλέ συχνέ μόνε με τα παιδιά του και δεν λαμβάνουν καν διατροφή ή μη οικονομική συνδρομή από του ε, συντρόφου. Και μάλιστα στο Βέλγιο έχουμε μια νομοθεσία όπου το κράτος κάνει μια προκαταβολή τέτοιες διατροφής και μετά το κράτος στρέφεται κατά του πατέρα που δεν ανέλαβε τις υποχρεώσεις, δεν πλήρωσε τη διατροφή αυτή. Νομίζω ότι χρειάζεται μια σαφής απάντηση και μια λύση για αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κακή οικονομική κατάσταση δεν θα πρέπει μόνο ένας γονιός να επιφορτίζεται την ευθύνη της ε, ανατροφής του παιδιού και της οικονομικής ευθύνης που αυτό συνεπάγεται. Μπορεί να μην απάντησα σε όλες. Περιμένω τις ανθρωπολογίες σας, θα τις εξετάσω προσεκτικά, θα προσπαθήσω είτε να τις ε, συγκεράσω, ε, για να μην αλλοιώσω και πολύ αυτή την έκθεση που την κρίνατε ως εξαιρετική και παραλαμβάνω τις ευχαριστήσεις μου. Ελπίζω ότι θα φτάσουμε στην Ολομέλεια με μια καλή έκθεση που θα βρήθει καλών προτάσεων και θα χαίρει και ευρεία συνένεση. Ευχαριστώ. Ε, ε, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ταραμπέλα. Για μια ακόμη φορά η αποδεικνύεται θα έλεγα η αφοσίωσή σας σε τέτοιου είδους θέματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις συναδέλφους για μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να κατεθάσουμε στην Ολομέλεια μια ενδιαφέρουσα έκθεση. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών η 7η Δεκεμβρίου 12η μεσημβρινή. Θα ψηφίσουμε την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου το απόγευμα και θα φτάσουμε ελπίζω στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του μηνός Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την συμμετοχή σας και για την παρουσίασή σας. Πηγαίνω τώρα στο επόμενο θέμα, το σημείο 7. Πρόκειται για την πλατφόρμα δράσης των Ηνωμένων Εθνών για την Ισότητα των Φύλων, Πεκίνο 15. Ενημερωτικά να πω ότι οι συντονιστές τον Οκτώβριο αποφάσισαν ότι η Επιτροπή μας θα διατυπώσει μια προφορική ερώτηση η οποία θα ακολουθηθεί από ψήφισμα. Ελπίζουμε να μπορέσει να γίνει δεκτή τον μήνα Φεβρουάριο για να προετοιμάσουμε την συνάντηση της Νέας Υόρκης στις αρχές Μαρτίου. Η Επιτροπή μας θα αποστείλει μια αντιπροσωπεία και μετά μάλιστα από τις σημερινές ανταλλαγές απόψεων γύρω από το θέμα της προφορικής ερώτησης Έχω πλέον την πρόταση της επιστολής την οποία θα στείλουμε ε, στα κράτη-μέλη, θα αντιλάβετε γύρω στις 10 Δεκεμβρίου. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών η 17η Δεκεμβρίου το απόγευμα. για να είμαστε σωστά επίκαιροι τώρα, σωστά ενημερωμένοι μάλλον για την συνάντηση αυτή, έχουμε και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος θα μας δώσει πληροφορίες για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Η Σουηδική Προεδρία δημοσίευσε μάλιστα πρόσφατα ένα έγγραφο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ασχολήθηκαν με το πρόγραμμα αυτό δράση στα διάφορα κράτη-μέλη. Έχει υπάρξει ενημέρωση προς τα κράτη-μέλη μέσω συγκεκριμένης ιστοσελίδας και δόθηκε και η δυνατότητα σχολιασμού γραπτά. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. θα μας ενημερώσει για το πού βρισκόμαστε σήμερα γύρω από το πρόγραμμα δράσης. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι η Μαρία Τομαζέτη θα σας κάνω μια παρουσίαση για το τι κάνουμε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη σχετικά με το πρόγραμμα δράσης του Πεκίνου και πώς προετοιμαζόμεθε για το λεγόμενο Πεκίνο συν 15. Να σας μεταφέρω ένα μικρό ιστορικό του, του έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Να σας πούμε τι συγκεκριμένα έχουμε κάνει επίσης για το Πεκίνο 15 και να σας πω πώς σκοπεύουμε να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Θεωρούμε ότι έχει σημασία ότι το Πεκίνο συν 15 θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και θα σας δώσω και κάποιες πληροφορίες για τη συνάντηση της Επιτροπής για την κατάσταση των γυναικών τον Μάρτιο του επόμενου έτους. Όπως γνωρίζετε έχουμε ξεκινήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την επεξεργασία δικτών και ποιοτικών και ποσοτικών για να παρακολουθήσουμε την πλατφόρμα δάσης του Πεκίνου ήδη από το 1999 και μετά. Αυτή ήταν μια απόφαση του Συμβουλίου και έχει υποστηριχθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπαθούμε να διατυπώσουμε δείκτες για πολλούς τομείς τους οποίους μας απασχολεί και μας ανησυχεί η κατάσταση. Έχουμε καλύψει σχεδόν όλους τους τομείς, με ελάχιστες εξαιρέσεις, για τη γυναίκα και τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, γυναίκα στην οικονομία, για συμφιλίωση και συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, για τις γυναίκες στην υγεία, για τις γυναίκες στους θεσμούς, γυναίκες και φτώχεια, γυναίκες και παιδιά και γυναίκες σε εμπόλεμες καταστάσεις. Ο τρόπος με τον οποίο δουλέψαμε μέχρι τώρα είναι μέσω συγκεκριμένων εκθέσεων που αναλύουν την κατάσταση στα κράτη-μέλη για να δούμε πού βρισκόμαστε και να δούμε πού έχουν υπάρξει βήματα πρόοδου. Μετά από τις πληροφορίες που πήραμε από τα κράτη-μέλη, προσπαθήσαμε να επιλέξουμε δείκτες αντιπροσωπευτικούς της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι ανά εξάμηνο, σχεδόν κάθε εξάμηνο, θα κατατίθενται οι εκθέσεις και τα συμπεράσματα σχετικά με τους τομείς που είπα μας ανησυχούν περισσότερο το 2005 ήταν καθοριστική στιγμή. Γιορτάσαμε τα 10 χρόνια του Πεκίνου 1. Η Λουξεμβουργιανή Προεδρία είχε προετοιμάσει μια έκθεση για το Πεκίνο συν 10 όπως λέγαμε τότε, εντοπίζοντας τους τομείς με τους οποίους θα έπρεπε να ασχοληθούμε. Βρισκόμαστε τώρα σε μια κρίσιμη στιγμή. Θα γιορτάσουμε του χρόνου την 15η κατά σειρά πλατφόρμα Προετοιμαζόμαστε με τη Φιλανδική Προεδρία, η οποία θα καταθέσει μία έκθεση που θα λαμβάνει υπόψη όλους τους δείκτες τους οποίους σταθήκαμε μέχρι τώρα, μεμονωμένα. Και στην ουσία θα υπάρξει μία ανακεφαλαίωση της κατάστασης στους τομείς όπου υπάρχουν ανησυχίες. Είναι μια ενδιαφέρουσα έκθεση, έχει γίνει αρκετά καλά αυτό δείχνει και τη συνεισφορά των διαδοχικών προεδριών αλλά και των κρατών μελών. Η Σουηδική Προεδρία συνεργάστηκε στενά με την Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών και αυτά τα οποία κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά κάποιο τρόπο έγιναν σε διάλογο θα έλεγα με την Περιφερειακή Επιτροπή του ΟΗΕ. Η έκθεση αυτή ανατομέα εντοπίζει τα προβλήματα, της προκλήσεις, τις πολιτικές τις οποίες πρέπει να υπάρξει παρέμβαση για την ισότητα των φύλων και για την εκλέπτυνση και βελτίωση των δικτών. Η έκθεση αυτή αποτελεί επίσης τη βάση για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που θα κατατεθούν κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας. Συμπτωματικά σήμερα θα πρέπει να γίνουν δεκτά τα συμπεράσματα αυτά. Περιλαμβάνουν τα βασικά μηνύματα στα οποία θα κινηθούμε στο μέλλον μας δίνουν την δυνατότητα να προχωρήσουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν Επιτροπή, σαν κρατημέλη, για να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την εφαρμογή της πλατφόρμας του Πεκίνου. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου εντοπίζουν κάποια κρίσιμα σημεία θα έλεγα κάτι το οποίο συζητήσαμε σήμερα και για την ισότητα των φίλων για τα στερεότυπα, τα σεξιστικά. Είναι κεντρικό πρόβλημα στα πλαίσια της προσπάθειας επίτευξης της ισότητας. Είναι μία από τις προτεραιότητες που έχει ήδη υπογραμμιστεί από το Προεδρείο, από το Συμβούλιο ενώ. Το mainstreaming δεν έχει ε, λειτουργήσει πλήρως όπως θα έπρεπε στον τομέα της ισότητας, δεν είναι δηλαδή μια πλήρης πραγματικότητα η ισότητα των ευκαιριών, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιτευχθεί και στον τομέα των μεταναστευτικών πολιτικών επίσης. Πρέπει να υπογραμμίσουμε επίσης τη σημασία που έχει η ισότητα των φύλων και στα πλαίσια της διαδικασίας της Λισαβόνας. Και όπως σας είπα, ασκείται μια κάποια κριτική σχετικά με τη διαθασιμότητα των δεδομένων. Δεδομένα έχουν βέβαια τα κράτη-μέλη σε, σε όλους τους τομείς που έχουν σχέση με το Πεκίνο, αλλά το θέμα είναι να τα συγκρίνει κανείς και να καταστήσει συμβατά σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτά τα δεδομένα. Και η διαδικασία προσπάθειας κατάρτισης των δικτών ναι με, ναι με λειτουργήσε σαν κίνητρο για τα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή στο μέλλον. Ένα άλλο κρίσιμο θέμα είναι ότι θα πρέπει στο μέλλον να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό με τον λεγόμενο διοικό τρόπο. Κίνητρα από τη μία και να μην ξεχνάμε ότι με το γενικό mainstreaming θα πρέπει να υπάρξουν και συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο την κατάργηση των διαφορών ανδρών γυναικών. Σχετικά με τη διαθεσιμότητα των δικτών και τον έλεγχο της προσπάθειας που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Οι υποδείξεις του Συμβουλίου είναι σαφείς. Καλεί το Συμβούλιο τα κράτη-μέλη με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεχίσουν να αναπτύσσουν δείκτες στους τομείς οι οποίοι δεν έχουν πλήρως καλυφθεί. Μία αναθεώρηση θα πρέπει να γίνεται με συστηματικό τρόπο στους τομείς στους οποίους υπάρχουν ήδη δείκτες και στο μέλλον θα πρέπει να προετοιμάσουμε ένα πρόγραμμα δράσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έχει ζητηθεί από το Συμβούλιο να κάνει ένα μεσοπρόθεσμο, μια μεσοπρόθεσμη έκθεση θα έλεγα απολογισμού. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ισότητα των ευκαιριών στον τομέα αυτό. Υπάρχει το θέμα βέβαια της τεχνικής δουλειάς η οποία θα πρέπει να γίνει στον τομέα του εκλεπτισμού, αν θέλετε, της εκλέπτυνσης μάλλον των δικτών και αυτή συνεχίζεται αλλά σε πιο συγκεκριμένες καταστάσεις γύρω από την 54η ε, συνάντηση της Επιτροπής για την Κατάσταση των Γυναικών προσπαθούμε να διαπιστώσουμε με ποιο τρόπο έχουμε συνεισφέρει στις εργασίες αυτής της συνάντησης. Αυτό έχει σημασία, γιατί όταν βρισκόμαστε σε ένα διεθνές πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παίζει πρωτοποριακό ρόλο σε σχέση με την πρόθεση των γυναικών. Πρόθεσή μας λοιπόν είναι να παρουσιάσουμε την έκθεσή μας αυτή σαν το ανώτατο σημείο της προσπάθειας την οποία έχουμε μέχρι τώρα κάνει. Και θα κάνουμε επίσης σε συνεργασία με την Προεδρία και κάποιες παράπλευρες εκδηλώσεις για να παρουσιάσουμε καλύτερα την έκθεσή μας αυτή και τη δράση μας Αυτά τα κάνουμε στα πλαίσια της συστηματικής προσπάθειας για συνέχεια των αποφάσεων στο Πεκίνο. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή και από τη Σουηδική Προεδρία. Η συνεργασία με την Προεδρία ήταν πολύ καλή μέχρι τώρα. και ακριβώς θα αναλάβουμε τον ρόλο της εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο CSW. Θα διοργανώσουμε και ένα φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών στις 4 και 5 Φεβρουαρίου και εκεί θα παρουσιάσουμε και τις θέσεις των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά. Αυτές είναι οι γενικές πληροφορίες που έχω να δώσω. Είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε να καταθέσετε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ε, για έναν τομέα που πραγματικά βρίσκεται στο επίκεντρο της ε, προσοχής μας. Πολύ σημαντικός ο τομέας για τις εργασίες και της Επιτροπής αλλά και για τη θέση των γυναικών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο σε αυτά. Αυτή η συνάντηση που θα λάβει η χώρα το Μάρτιο στη Νέα Υόρκη θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και είμαι πεπισμένη ότι οι συνάδελφοί μου στην Επιτροπή επιθυμούν ε, διακαώς ε, η Επιτροπή μας ε, να παρουσιαστεί ως Επιτροπή Ψηλού Κύρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταστεί απόλυτα σαφές το τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέρουμε μεγάλη ευθύνη για την Νέα Υόρκη. Πάνω σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε όλες αυτές τις πληροφορίες που ήταν και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Είναι πολύ σημαντικό το Συμβούλιο να εγκρίνει αυτά τα συμπεράσματα και ελπίζω ε, να μπορείτε και εσείς κάποια στιγμή να μας πείτε κατά πόσον πράγματι τα ε, συμπεράσματα αυτά εγκρίθηκαν ή όχι. Επιτρέψτε μου να κάνω και εγώ κάποιες ε, παρατηρήσεις αυτά που είπατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που το θέμα των στερεοτύπων σχετικά με τα δύο φύλλα θα έχει ε, ψηλή προτεραιότητα. Γιατί νομίζω από εκεί, από αυτά τα στερεότυπα, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό το επάγγελμα που διαλέγουν οι άνδρες και οι γυναίκες. Το να υπάρχει σωστή αντιμετώπιση βαδίζουμε στο σωστό δρόμο. Όσον αφορά τώρα την ε, διάσταση του φύλου σε πάρα πολλούς τομείς, ε, το mainstreaming και εγώ προσωπικά δεν είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι το mainstreaming streaming, αυτή η διάσταση του φύλου μόνη της μπορεί να επιφέρει πολλά πράγματα. Πρέπει να συνδυαστεί και με άλλα μέτρα, συγκεκριμένα μέτρα. Όσον αφορά τώρα τη στρατηγική της Λισαβόνας και εγώ θεωρώ ότι ο τομέας αυτός είναι πολύ σημαντικός και εμείς στην Επιτροπή μας ασχολούμεθα σε βάθος με αυτή τη στρατηγική γιατί όλα αυτά τα θέματα έχουν σχέση με την ισότητα των δύο φύλων. Και τέλος μια παρατήρηση θα μου επιτρέψετε σχετικά με την διαθεσιμότητα συγκρίσιμων στατιστικών από τα κράτη-μέλη. Βεβαίως είναι κομβική σημασία όταν συζητάμε για θέματα ισότητας των δύο να έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά τα χρειαζόμαστε έτσι ώστε οι θέσεις μας να μην είναι ε, απαραίτητα ε, ισχυρισμοί, αλλά να τεκμηριώνονται και με ε, συγκεκριμένα στοιχεία. Για μένα λοιπόν αυτό σχετίζεται άμεσα και με τη δουλειά αυτή του Ινστιτούτου περί των δύο φύλων. Αυτό το Ινστιτούτο πρέπει εδώ να δραστηριοποιηθεί. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα πολύ σημαντικό που πρέπει να το εξετάσει η Επιτροπή μας. Τι είναι αυτό το Ινστιτούτο των δύο φύλων και ποιο ακριβώς είναι το έργο του. Αυτά είχα να πω εν συντομία. Ε, τα σχόλια τα δικά μου και τώρα ξεκινάει η συζήτηση και οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν παρακαλώ μπορούν να λάβουν το λόγο. Ευχαριστώ. Διάβασα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου μία σύσταση προς τα κράτη-μέλη ως προς την υιοθέτηση μέτρων που θα επιτρέπει στους άνδρες και στα αγόρια να αναλαμβάνουν τμήμα των οικογενειακών ευθυνών ισότιμα με τις γυναίκες. Πολύ ωραία όλα αυτά. Γιατί όμω το Συμβούλιο δεν θέλει να υποστηρίξει την έκθεση κυρίας Εστρέλα που ζητά θέσπιση της άδειας πατρότητας. Αυτό δεν είναι αντίφαση. Ehm, Καλώς, η κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ. Μία παρατήρηση ως προς το προηγούμενο σχόλιο. Η έκθεση αστρέλα δεν υπάρχει. Οπότε ούτε το Συμβούλιο ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να την ε, υποστηρίξουν. Ελπίζω η πρόταση που θα υποβάλουμε είναι πολύ πιο υπεύθυνη από αυτή που εξετάζεται τώρα για να μας πάρουν πραγματικά στα σοβαρά και για να προωθήσουμε την προστασία της μητρότητας γιατί αυτό είναι τελικά ο στόχος αυτής της πρότασης ε, μεταρρύθμισης. Τώρα για το Πεκίνο συν 15. Ήμουν στο Πεκίνο, ήμουν και στο Πεκίνο συν 5. Και τότε ήταν και η Λουξεμβουργιανή Προεδρία το 1985. Ήμουν και στη συνδιάσκεψη της Κένιας. Και είναι σαφές ότι όλα τα σχετικά με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την ισότητα θα γίνουν θα τα διαχειριστεί η Προεδρία και θα εξασφαλίσει και το συντονιστικό ρόλο. Δηλαδή δεν είναι οι εθνικές αντιπροσωπείες που θα διαχειριστούν αυτά τα θέματα, αλλά η Επιτροπή. Αυτή θα είναι η συντονίστρια. Και πραγματικά είναι πολύ δύσκολος αυτός ο ρόλος. Το θυμάμαι στην Κένια. Τώρα ίσως στο Πεκίνο συν 15 τα πράγματα δεν είναι τόσο φιλεγόμενα όσο στην Κένια. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να υπάρξει μια πειθαρχία μεταξύ των χωρών μέλλον είχα τεράστιο πρόβλημα να επιβάλλω κάποια πειθαρχία λέγοντας ότι δεν θα έπρεπε τα κράτη-μέλη μεμονωμένα να λάβουν το λόγο, αλλά η Προεδρία εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω όμως ότι τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα για το στην 15. Και εκεί θα μπορούσαμε να πάμε και να γίνουμε και υπόδειγμα συμπεριφοράς δίνοντα το καλό παράδειγμα και λέγοντα ότι η δική μα πολιτική ισότητα φίλων και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών είναι απαράμιλη. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο. Να μην ε, διαρριγνύουμε συνέχεια τα ημάτια μας και να παραπονιόμαστε και να συμπληρούμε ότι η πολιτική μας επιδέχεται βελτιώσεις. Σίγουρα ε, βελτιώσεις χρειάζονται, αλλά ως προς την εφαρμογή περισσότερο, όχι ως προς τη σύλληψη. Πιστεύω ότι μπορούμε να γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση. Και μπορούμε να πάμε και στο Πεκίνο στις 15 και στη Νέα Υόρκη με υπερηφάνεια για ό,τι έχουμε ήδη επιτύχει. Και πολλές διεθνείς οργανώσεις και οργανώσεις δικαιωμάτων προστασίας των γυναικών. Δεν θα πρέπει λοιπόν ε, να αφήσουμε να μας επισκιάσουν. Πρέπει στη Νέα Υόρκη να καταδείξουμε εμείς τον δρόμο και να μεριμνήσουμε έτσι ώστε άλλοι να ακολουθήσουν το δικό μας το καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ. Ortega. Your micro. You. you it's okay. It No, switch it on. Då går ordet till ehm, kommissionen. Πρόεδρος, η εκπρόσωπος της ε, Κομισιόν θα λάβει για άλλη μια φορά το λόγο, αλλά πρώτα η κυρία Τομασέτη, μισό λεπτό, αν έχει την καλοσύνη, Άλλη μία συνάδελφος ε, θέλει να λάβει το λόγο, η κυρία Κλάς. Κυρία Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να σας πω άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ε, παρουσίαση της ε, Κομισιόν και θέλω να σας πω το εξής. Εγώ ήμουν στη Νέα Υόρκη για την εκδήλωση Πεκίνου στην 5 και σκέφτηκα το εξής. Πού είναι κάτι το χειροπιαστό επιτέλους. Δεν θα πρέπει να κάνουμε το λάθος ε, οτιδήποτε σημαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο να το συμπεριλάβουμε σε μία έκθεση, σε ένα χοντρό τόμο που κανείς θα διαβάσει. Θα πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε να έχουμε αν θέλετε ε, κάποιο κεντρικό μήνυμα. Εγώ δεν το ξέρω αυτό, αλλά έχουμε ακόμα χρόνο και μπορούμε να το σκεφτούμε. Και ακόμα και ο τίτλο συν 5, συν 10, συν 15. Νομίζω ότι σιγά σιγά ε, θα πρέπει να βρούμε κάποια άλλη μορφή διατύπωσης που να τραβάει περισσότερο την προσοχή. Και όχι απλά να λέμε 5, συν 5, συν 10, 15. Ε, θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να προσέξουμε να εκφραστούμε με μεγαλύτερη σαφήνεια γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία νομίζω ότι μπορούμε να συνδέσουμε. Ευχαριστούμε κυρία Κλάς. Νομίζω ότι αυτή ήταν και μία έκκληση προς την Πρόεδρο και τους συντονιστές που θα κάνουν αυτή την προφορική επερώτηση μετά το ψήφισμα. Τα συγκρατήσαμε λοιπόν όλα αυτά. Από ό,τι φαίνεται κανείς άλλος συνάδελφος δεν επιθυμεί να λάβει το λόγο. Ως εκ τούτου θα μου επιτρέψετε να ξαναδώσω το λόγο στην Κομισιόν. Η κυρία Τομασέτη έχει το λόγο. Ε, thank you very much. Ε, it's just to, uh, σας ευχαριστώ. Η Προεδρία θα εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά και τα κράτη-μέλη και είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να σταθεί σαν υπόδειγμα γιατί έχουν πράγματι υπάρξει πρόοδος και η έκθεση που προετοίμασε η Σουηδική Προεδρία δείχνει ποια είναι αυτή η πρόοδος και ποιες είναι και οι δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας και στα πλαίσια αυτά τα διεθνή. Θα φανεί ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω πρόοδου. Πολλές χώρες θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται της προσπάθειας αυτής γιατί σίγουρα υπάρχει πολλή εμπειρία ο συντονισμός είναι κάτι το αρκετά δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Νομίζω ότι μέχρι τώρα εμπειρίες δείχνουν ότι μπορούμε να πετύχουμε καλά σχετικά αποτελέσματα. Θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα προσπαθούν να εκπροσωπήσουν τις αξίες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε. Οι συντονιστές λοιπόν και το Προεδρείο θα καταθέσουν μια προφορική ερώτηση όπως είπαμε και θα ακολουθήσει ένα ψήφισμα. Ήδη ακούσαμε το χρονοδιάγραμμα. Εγκαταλείπουμε λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα για το Πεκίνο 15, τουλάχιστον για σήμερα. Θα έχουμε τη δυνατότητα όμως στο μέλλον να επανέλθουμε. Υπάρχει ένα επιπλέον θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σήμερα, αφορά τη διαφορά αμοιβή. Είναι ένα θέμα το οποίο γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι. Είδαμε ότι το θέμα αυτό παραμένει σε εκκρεμότητα. Η Επιτροπή στις 3 Μαρτίου ξεκίνησε μια εκστρατεία πληροφόρησης Η κυρία Μπάουερ το 2008 συνέταξε μια έκθεση γύρω από το θέμα αυτό που έγινε δεκτή το Νοέμβριο η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μαζί μας σήμερα και θα μας ενημερώσουν για την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η Επιτροπή. Έχετε το λόγο κυρία Μπανκέα. Ελπίζω να μην κάνω λάθος το όνομα για μια ακόμη φορά. Σας καλωσορίζω και σας ακούμε με ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και σας ε, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας ε, παρουσιάσω την εκστρατεία ενημέρωσης ε, και συνειδητοποίησης ε, σχετικά με την διαφορά στην αμοιβή, διαφορά αμοιβής. Θα ήθελα λοιπόν με την παρουσίασή μου αυτή να σας κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή ε, σε αυτό το θέμα που είμαι σίγουρη ότι το γνωρίζετε πολύ καλά αλλά παρόλα αυτά ε, θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να σας πω τι είναι ακριβώς αυτό να σας δώσω και τα τελευταία στοιχεία και μετά θα ήθελα να σας δείξω τι ακριβώς ε, κάναμε κατά τη διάρκεια της εξτρατείας μας για τη διαφορά αμοιβή. Πρώτα απ' όλα, τι είναι η διαφορά αμοιβή. Η διαφορά αμοιβή είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που κερδίζουν οι άνδρες και αυτό που κερδίζουν οι γυναίκες. Αυτή τη στιγμή ε, σε αριθμούς μιλάμε για ένα περίπου 17,4% είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που με εντυπωσιάζει ε, σχετικά με το θέμα αυτό, με την αμοιβή, τη διαφορετική αμοιβή, αν δούμε λιγάκι πώς εξελίσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα διαπιστώσουμε ότι επιμένει η διαφορά και σε ορισμένα κράτη-μέλη μάλιστα διευρύνεται. Άρα δηλαδή Μιλάμε για ένα δύσκολο να αντιμετωπιστεί φαινόμενο. Και βεβαίως αυτό το χάσμα ανησυχεί και κάτω από το πρίσμα της ισότητας, αλλά και κάτω από το πρίσμα του να διασφαλιστεί η ανάπτυξη και η θέση εργασίας στην Ευρώπη. Γιατί λοιπόν υπάρχει και επιμένει αυτή η διαφορά. Κάποιοι κάποτε είπαν ότι αυτή η διαφορά αντικατοπτρίζουν όλες τις διαφορές ε, τις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας. Είναι ένα πολύ περίπλοκο φαινόμενο και για να αντιμετωπιστεί νομίζω ότι πρέπει κανείς ε, να κατανοήσει και τα αίτια που οδηγούν σε αυτό. Πρώτα απ' όλα λοιπόν έχουμε ως αίτιο την ε, διακριτική μεταχείριση. Βεβαίως ε, αυτή η μεταχείριση σιγά σιγά ε, εκλείπει, δηλαδή η διακριτική μεταχείριση δεν είναι πλέον τόσο άμεση γιατί έχει γίνει περισσότερο ε, εξελιγμένη η φέρπουσα θα τη χαρακτήριζα. Είναι λοιπόν δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Εξάλλου η διαφορά στην αμοιβή έχει και άμεση σχέση με την αξία που αποδίδει μια κοινωνία και οι εργοδότες ε, ε, στην γυναική εργασία σε αντίθεση με την ανδρική. Εξάλλου υπάρχει και ένα θέμα ε, διαφοροποίησης στην αγορά εργασίας όπου εκεί έχουμε τομείς που εξακολουθούν να είναι χαρακτηριστικά γυναικοί σε αντίθεση με αυτούς που είναι χαρακτηριστικά ανδρικοί. Εξάλλου, αυτό το, αυτή η διαφορά έχει, όπως σας είπα, άμεσα σχέση με τα στερότυπα και με τις επιλογές των ανδρών και των γυναικών όταν επιλέγουν κάποια επαγγέλματα. Η διαφορά στην αμοιβή έχει και άμεση σχέση με τις ε, δυσκολίες ε, συμφιλίωσης ε, μιας ε, επαγγελματικής δραστηριότητας με την οικογένεια και την ε, ιδιωτική ζωή των ανθρώπων. Εξάλλου η διαφορά αυτή σχετίζεται και με φαινόμενα που θα τα χαρακτήριζα αυθαίρετα. Όλα αυτά λοιπόν μας δείχνουν ότι είναι ένα πολύ περίπλοκο φαινόμενο, το οποίο όπως σας είπα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, ακριβώς γιατί είναι περίπλοκο. Οι συνέπειες ε, αυτής της ε, διαφοράς είναι πρώτα απ' όλα ε, διασπάθηση πόρων για το σύνολο της οικοσομίας. Χάνονται ταλέντα που θα μπορούσαν να φέρουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας και για τους εργοδότες τους και επίσης αυτό το, αυτή η διαφορά έχει αρνητικές επιπτώσεις ε, στην ε, οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών. Εξάλλου επηρεάζει και τη φτώχεια κυρίως ε, όταν έχει κανείς κατά νου τις ανήπαντρες μητέρες στην αγορά εργασίας. Ας πάμε τώρα λίγο στα στοιχεία. Σας έχω φέρει μαζί μου τα στοιχεία για κάθε κράτος μέλος και για το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αυτή τη στιγμή ενέρχεται σε 17,4%. Ε, πρόσφατα άλλαξε η μέθοδος ε, ε, βελτιώθηκε ο υπολογισμός αυτής της διαφοράς και εδώ στο γράφημα βλέπετε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα κράτη-μέλη, ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Δηλαδή υπάρχουν κράτη-μέλη όπου η διαφορά είναι ε, μικρότερη από 5% αλλά έχουμε και άλλα όπου η διαφορά ξεπερνάει το 30%. Βλέποντας λοιπόν αυτά τα στοιχεία διαπιστώνουμε ότι ε, υπάρχουν τρεις ομάδες χωρών. Μία ομάδα χωρών όπου αν πάρει κανείς ε, το κάτω μέρος του γραφήματος, εκεί εντάσσονται Ιταλία, η Μάλτα, η Πολωνία, εκεί η διαφορά στην αμοιβή είναι αρκετά μικρή. Δηλαδή αυτό δεν σημαίνει ότι στη Μάλτα, την Ιταλία και την Πολωνία ε, όλα βαίνουν καλώς όσον αφορά την θέση των γυναικών στην αγορά εργασία. Όχι, εδώ η διαφορά αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η απασχολησιμότητα των γυναικών σε αυτές τις χώρες είναι πολύ περιορισμένη. Σε αυτές λοιπόν τις ε, χώρες οι γυναίκες που δεν έχουν πολλά προσόντα μάλλον δεν απασχολούνται και γι' αυτό όπως σας είπα και η διαφορά στις χώρες αυτές είναι σχετικά μικρή. Υπάρχει και μία άλλη ομάδα χωρών όπου η αγορά εργασίας είναι πολύ επιλεκτική και διαφοροποιημένη. Κύπρος, Εστονία, Σλοβακία, Φινλανδία. Εκεί ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η έντονη διαφοροποίηση, η διαφορά ε, στην αγορά εργασίας, ε, στην αμοιβή μάλλον, είναι πολύ έντονη. Εδώ έχουμε πολλές γυναίκες που απασχολούνται άλλη ομάδα τώρα. Γυναίκε, ομάδε χωρών, όπου γυναίκε απασχολούνται με ορική απασχόληση. Ε, Ολλανδία, Αυστρία, Γερμανία και εκεί ε, ο ξεπερνάει, ναι, ξεπερνάει διαφορά το μέσο όρο. Ποια είναι τα μέτρα που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσει αυτό το μισθολογικό χάσμα Υπάρχουν αναμορφωτικέ διατάξεις για τις αμοιβέ. Και μάλιστα πέρυσι ορτάσαμε την πέτειο από τη Συνθήκη της Ρώμης και την πρώτη διάταξη για την ισότητα των δύο φύλων, που ήταν η διάταξη ίση αμοιβή για ίση εργασία. Και μάλιστα η διάταξη αυτή στη συνέχεια ε, μετατράπηκε σε μια οδηγία του ε, το 57 για την, το 57 συγγνώμη, για την ισότητα αμοιβή και στη συνέχεια επεξεργαστήκαμε αυτές τις αρχές ε, της ίσης αμοιβή για ίση εργασία και μετά είπαμε ε, ίση αμοιβή για ίση εργασία και εργασία ίσης αξίας και είχαμε και άλλες ε, οδηγίες του 2002 και την αναδιατύπωση την πρόσφατη αναδιατύπωση της οδηγίας ε, που κατοχύρωνε και πάλι αυτές τις αρχές. Κατά τη γνώμη μου, Υπάρχει αυτή τη στιγμή κοινωτική νομοθεσία και μάλιστα αρκετά περιεκτική για το θέμα της ισότητας των αμοιβών. Και είχαμε και πολλές προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για θέματα ισότητας αμοιβών. Και εκεί ήταν σημαντική νομολογία του ΔΕΚ σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και την ερμηνεία των εφισταμένων διατάξεων για την ισότητα αμοιβών. Γιατί το ΔΕΚ υιοθέτησε πολύ διασταλτική ερμηνεία και πολύ γενναιόδορη ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων για την ισότητα των αμοιβών. Έχουμε λοιπόν και περιεκτική και εκτεταμένη νομοθεσία, αλλά και εκτεταμένη νομολογία του ΔΕΚ για το θέμα της ισότητας των αμοιβών. Αλλά δεν έχουμε μόνο νομοθετικές διατάξεις, έχουμε και το θέμα της ισότητας των αμοιβών ως προτεραιότητα στον οδικό χάρτη για την ισότητα των φύλων και μάλιστα η διάμεση στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων αναφέρει το θέμα της διαφοράς της αμοιβή. Η ισότητα της αμοιβή είναι μία από τις τέσσερις προτεραιότητες της πολιτικής μας για τη ισότητα των φύλων. Έχουμε ε, την οικονομική ανεξαρτησία των ανδρών και των γυναικών, την, ε, το συνδυασμό επαγγελματική και οικογενειακή ζωή, η πρόθεση τη ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψη αποφάσεω και στην κατάργηση των ε, στερεοτύπων. Και τέσσερι τέσσερις αυτούς τομεί, το θέμα τη ισότητας των αμοιβών λαμβάνεται υπόψη. Το 2007 υιοθετήσαμε μια ανακοίνωση για τη γεφύρωση αυτού του μισθολογικού χάσματος και προτείναμε συγκεκριμένες δράσεις. Μία από αυτές ε, που περιλαμβανόταν στην ανακοίνωση ήταν η ενημερωτική εκστρατεία για το θέμα αυτό, που θα σας παρουσιάσω λίγο αργότερα. Εκτός όμως από τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγιναν και πολλές συζητήσεις για την ισότητα των αμοιβών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχαμε και ένα νομοθετικό ψήφισμα πρόσφατα της κυρίας Μπάουερ, πολύ ενδιαφέρον, με πολλές και ενδιαφέρουσες και εύστοχες προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του μισθολογικού χάσματος. Έχουμε και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο της ισότητα των φύλων που έθεσαν τα κράτη-μέλη και το πλαίσιο δράσεων των κοινωνικών εταίρων που προσπαθεί να αντιμετωπίσει και πάλι αυτή τη διαφορά αμοιβή. Και επανέρχομαι στο θέμα της ενημερωτικής εκστρατείας. Ξεκίνησε η ενημερωτική εκστρατεία και εκστρατεία φύπνιση στο Μάρτιο του 2009 με στόχο την αφύπνιση, τη συνειδητοποίηση αυτού του προβλήματος και Απόδεκτης ε, η κοινός στόχο, ακροτήριος στόχος ήταν ε, οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι πολίτες και φυσικά το βασικό μήνυμα της ε, ενημερωτικής εκστρατείας είναι η γεφύρωση αυτού του μισθολογικού χάσματος, η μείωση αυτής της διαφοράς αμοιβή και τονίζουμε και τα ωφέλη που απορρέουν από μια τέτοια κατάργηση αυτής της διαφοράς. Θα έχουμε πολλά κοινωνικά ωφέλη από αυτή την απάλληψη της διαφοράς αμοιβή και για την οικονομία αλλά και για τους εργαζόμενους. Εγκαινιάσαμε αυτή την ε, εκστρατεία με εκδηλώσεις ε, που προβλήθηκαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο Επίτροπος Σπίτλα έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη τύπου το Μάρτιο και μάλιστα διοργανώσαμε και ένα σεμινάριο όπου ενημερώσαμε δημοσιογράφους και τους δώσαμε και πολλά στοιχεία την προσπάθεια αυτή κατά πολέμηση της διαφοράς αμοιβής. Ήταν πολύ επιτυχημένο αυτό το σεμινάριο των δημοσιογράφων γιατί έτσι προβλήθηκε το θέμα αυτό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκτεταμένα. Μάλιστα είχαμε και τον ιστότοπο σε 22 γλώσσες με εκτεταμένες πληροφορίες για τη διαφορά αμοιβών. Είχαμε και σύντομα βίντεο κλιπ για το θέμα της διαφοράς αμοιβής. Και μάλιστα συνοδεύσαμε την εκστρατεία μας με διάφορες φωτογραφίες, εικόνες και μηνύματα ξεκινώντας από τα παιδιά και φτάνοντας στους ενήλικες. Προσπαθήσαμε να δείξουμε, να δείξουμε τη σημασία της διαφοράς της αμοιβή σε τέσσερα στάδια της ζωής των ανδρών και των γυναικών. Ξεκινήσαμε με τα βρέφη, δείχνοντας ότι τα στερεότυπα ξεκινούν από πολύ νωρίς ε, στην ζωή του ανθρώπου από τη βρεφική ηλικία και οι επιλογές που κάνουν για τη σταδιοδρομία του οι νέοι έχουν σχέση με το φίλο τους. Μετά δίνουμε τις φωτογραφίες 2-30 ε, χρονών και εκεί μιλούμε για την αξία της εργασίας. Την αξία της εργασίας των γυναικών ε, έναντι της αξίας της εργασίας των ανδρών. Και για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο ότι το φύλλο επηρεάζει μερικές φορές τις επαγγελματικέ επιλογές, ε, λέμε ότι το 59% των αποφύτων πανεπιστημίου σήμερα είναι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, σε πολλές, ε, σε πολλές ε, κατευθύνσεις σπουδών υπερέχουν οι άνδρες. Δίνω μετά τη φωτογραφία μιας οικογένειας, ενός ζευγαριού με ένα παιδάκι, Κάποτε ο πρώην Σουηδός διαμεσολαβητής είπε ότι όταν ε, δύο σύζυγοι αποκτούν παιδί, ε, διευρύνεται το μισθολογικό χάσμα. Και αυτό μας λένε οι στατιστικές, ότι οι γυναίκες που έχουν παιδιά, τη στιγμή μάλλον που αποκτούν παιδί, δημιουργείται μια καμπή στην ε, επαγγελματική τους δραστηριότητα και εκεί αρχίζει και διευρύνεται η διαφορά αμοιβή ε, υπέρ του ανδρός. Και μάλιστα αυτό επηρεάζει και το ποσοστό απασχόληση των ανδρών. Ε, οι άνδρες με παιδιά εργάζονται κατά ποστό 91% ενώ οι γυναίκες με παιδιά εργάζονται σε πολύ μικρότερο βαθμό. Μόνο 62% των γυναικών που έχουν παιδιά εργάζονται σε αντίθεση με το 91% των ανδρών. Και αυτό δείχνει το χάσμα που δημιουργείται και που διευρύνεται με την απόκτηση των παιδιών, με την έλευση των παιδιών στην οικογένεια. Βέβαια και η μερική απασχόληση, όπως ξέρετε, ασκείται κατά κανόνα από τις γυναίκες. Πάνω τα τρία τέταρτα της μερικής απασχόλησης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, γίνεται από γυναίκες. Έχουμε την τελευταία φωτογραφία δύο συνταξιούχων για να δείξουμε ότι η συσσόρευση της, χαμηλότερης, ε, της χαμηλής αμοιβή ε, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής έχει επίδραση και στο ύψος της σύνταξης. Δείχνουμε από τη φωτογραφία αυτή ότι ο κίνδυνος φτώχειας στις γυναίκες συνταξιούχες είναι πολύ ψηλότερος από τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι άνδρες. Και Αυτά τα στοιχεία μοιράσαμε στα γραφεία μας στις χώρες μέλη, δώσαμε και φυλάδια, ένα χάρτη της Ευρώπης με τις μισθολογικές διαφορές, επαναλαμβάνω κάποια, κάποιες μικρές σύντομες βιντεοτενίες, βιντεοκλίπ. Επίσης είχαμε και άλλο υλικό που το μοιράσαμε στις διάφορες εκδηλώσεις που οργανώσαμε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το πιο πρωτότυπο ήταν ε, ένα υπολογιστή που μοιράσαμε, ένα κομπιουτεράκι για να μπορεί να υπολογίζει κανείς εύκολα τη διαφορά μισθών. Είχαμε και έναν ιστότοπο, δημιουργήσαμε και έναν ιστότοπο με πληροφορίες για τις διαφορές ε, στις αμοιβέ, που όπως σας είπα μεταφράστηκε σε 22 γλώσσες και με γραφεία και σημεία επαφή ε, και links σε όλα τα κράτη-μέλη για να μπορεί κανείς να ευθύνεται εκεί και να λαμβάνει πληροφορίες. Είχαμε και οπτικοακουστικά μέσα και σύντομα βιντεάκια που μπορείτε να τα κοιτάξετε επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα. Τώρα, γιατί έχει σημασία το είπα και τελειώνω με κάποιες φωτογραφίες που δείξαμε και στα μέσα ενημέρωσης ε, στα κρατημέλη αλλά και με αφήσει που αναρτήσαμε σε, στις έδρες των κοινοβουλίων αλλά και σε λεωφορεία σε διάφορες ε, πόλεις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αυτές ήταν οι γαντοαφήσεις στον Μπελιάρ, ε, στη Γέφυρα, δεν ξέρω αν τα, τα προσέξατε αυτό το Μάρτιο. χρησιμοποίησαμε και εφημερίδες για διαφημιστικούς λόγους. Εδώ φαίνονται οι πόλεις στις οποίες των οποίων τα λοφορεία χρησιμοποιήσαμε σαν πλατφόρμες για διαφήμιση. <clears throat> Πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Χρησιμοποιήσαμε επίσης αυτό το υλικό εκστρατεία σε διάφορα στάντ, περίπτερα, στα πλαίσια της προσπάθειας ΣΕΡΚΟΣ που χρησιμοποιεί η Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση σε πολλές πόλεις της Ευρώπης, δίνοντας πληροφορίες για το τι κάνει η Ευρώπη στον κοινωνικό τομέα. Η δεύτερη φάση της εκστρατείας προβλέπεται για το 2010 τρεις βασικές δραστηριότητες, εταιρική σχέση, οικοδόμηση εταιρική σχέση σε όλα τα κράτη-μέλη. Βασιζόμαστε στις εμπειρίες τις οποίες αποκτήσαμε στην πρώτη περίοδο της εκστρατείας. 50 με 100 εταίροι σε πολλά κράτη-μέλη θα λειτουργήσουν σαν πολλαπλασιαστές θα έλεγα της ε, προσπάθειας πληροφόρησης. Ένα δεύτερο βήμα είναι τα μέσα ενημέρωσης με πιο αποκεντρωμένο τρόπο από ότι στην πρώτη φάση. Θα διαφημίσουμε την προσπάθεια και σε τοπικές εφημερίδες, στα δημόσια μέσα μεταφορών, λεωφορεία, αεροπλάνα, σιωδρομικούς σταθμούς. Ε, τα αεροδρόμια θα χρησιμοποιήσουμε τα των πρωτεύουσών, ενώ σιωδρομικούς σταθμούς θα χρησιμοποιήσουμε μικρότερες πόλεις. Αυτό θα το κάνουμε γύρω στο μήνα Μάρτιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επηρεάσουμε καλύτερα τις συναντήσεις. Τελειώνοντας, εδώ έχετε τη διεύθυνση του ιστοτόπου μας. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περαιτέρω ερωτήσεις. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ. Ε, πρόκειτο για ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές ε, που μόλις κατετέθησαν θα σας διανεμηθούν και θα συνεχίσετε την ε, μελέτη τους αν θέλετε με το δικό σας ρυθμό. Λίγα λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. Ίσως κάποιες πολύ σύντομες ερωτήσεις ο κύριος Ταραμπέλα, ο Βίρ και Τόμσον μετά. Αλλά μόνο σύντομες, σύντομα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια αυτή ενημέρωσης μέσω διαφημιστικών σημείων. Μήπως θα μπορούσε να υπάρξει και μια δυνατότητα αρνητικής ενημέρωσης. Αυτή είναι μια θετική προσπάθεια την οποία κάνουμε. Οι ιδιωτικέ επιχειρήσεις όμως και ιδιαίτερα οι μεγάλες πολυεθνικές οι οποίες πρέπει να κάνουν τη μεγαλύτερη προσπάθεια σε επίπεδο στελεχών κτλ. Μήπως θα μπορούσαμε αρνητικά να κατονομάζουμε ας πούμε τις επιχειρήσεις αυτές που έχουν διαφορετικές αμοιβέ για γυναίκες και για άνδρες, διαφορετικά ποσοστά γυναικών σε επίπεδο διευθυντικών θέσεων. Γνωρίζω ότι ουσιαστικά όλοι λέγουν ότι είναι ευαίσθητοι σε σχέση με την εικόνα τους και πολλές επιχειρήσεις θα θελήσουν να αποφύγουν αυτή την αρνητική εικόνα και θα πρέπει να λειτουργήσει θετικά για τις γυναίκες. Καλώς. Παρακαλώ σύντομες οι ερωτήσεις, όχι πάνω από ένα λεπτό, κυρία Όβιρ. Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Η κατάσταση δυστυχώς δεν έχει βελτιωθεί. Σε κάποιες χώρες γίνονται βήματα προόδου, σε άλλες χώρες όμως τα πράγματα χειροτερεύουν. Και αυτό ισχύει για τη δική μου χώρα, την Εσθονία. Λυπάμαι για αυτή την εξέλιξη, ντρέπομαι για αυτή την εξέλιξη. Και διαρωτώ με αν η εκστρατεία που κάνατε στη Βουδαπέστη, στην Πολωνία, Ξέρετε ότι έχουν διαφορές στις αμοιβέ 20% στην Πολωνία, 30% στην ε, Εστονία. Κάνατε προσπάθειες και σε χώρες όμως όπου η διαφορά στις αμοιβέ δεν είναι πολύ μεγάλη. Γιατί δεν διαλέξατε τις χειρότερες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και ε, από ό,τι κατάλαβα έγινε λόγος και για την προώθηση των γυναικών. Δηλαδή στην οδηγία δεν ασχολούμεθα μόνο με τη διαφορά στην αμοιβή αλλά και με τις, ε, ε τη σταδιοδρομία των γυναικών. Εμείς στη Walmart το 2007 σε αυτό το μεγάλο ε, κατάστημα επενέβησαν τα συνδικάτα και καταδικάστηκε, επιβλήθηκε τελικά στο σούπερ μάρκετ ένα σημαντικό πρόστιμο γιατί το σούπερ μάρκετ δεν είχε ε, προβιβάσει τις γυναίκες ε, όπως και τους άντρες. Νομίζω λοιπόν εμείς ε, στην Ευρώπη δεν ασχολούμεθα με τη σταδιοδρομία των γυναικών. Αυτό όμως είναι ένα σημαντικό στοιχείο στη διαφορά στην αμοιβή και θα ήθελα να γνωρίζω ε, ποια είναι ακριβώς η άποψη των γυναικών σχετικά με αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ κύριε Λούλινγκ για ένα λεπτό και μετά κυρία Μπάουερ. Καταρχήν, μία αντίδραση σε αυτά που είπε προλαλήσασα. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε νομοθεσία για την ε, η συμμεταχείριση ε, για τις προαγωγές από το 1996 υπάρχει τέτοια νομοθεσία και πρόσφατα αναθεωρήθηκε. Και περιμένω με ανυπομονησία την έκθεση αυτή για να την αναλύσουμε διεξοδικά. Έμεινε εμβρόντιτη από το γεγονός ότι η Μάλτα που είναι πρωταθλήτρια με, το, με τη χαμηλότερη μισθολογική διαφορά αναφέρεται στον κατάλογο. Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί όμως. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τον κατάλογο αυτό όπου έχουμε τα στατιστικά γιατί στην Μάλτα δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο το ποσοστό γενικών που εργάζεται. Προσοχή λοιπόν στην ανάλυση και μερικές φορές τα στατιστικά στοιχεία παρά είναι γενικά. Η κυρία Τόμσον είπα, μια και έχουμε νομοθεσία, θα πρέπει να προωθήσουμε τις γυναίκες ε, και να τις προαγάγουμε περισσότερο όπως γίνεται και με τους άνδρες. Έχουμε την νομοθεσία, αλλά δεν την εφαρμόζουμε καλά. Δεν θέλω συζήτηση τώρα, μόνο ολιγόλεπτες ερωτήσεις για να ακούσουμε, προλάβουμε να ακούσουμε και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Μπάουερ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Τρεις ερωτήσεις. Κοιτάξτε, πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Εδώ μιλάμε για, τον, για το ρομίστιο. Και όταν λέμε ότι η διαφορά είναι μεγαλύτερη στην αμοιβή γιατί είναι περισσότερες οι γυναίκες που εργάζονται με μερική απασχόληση. Αυτό δεν ισχύει. Ε, στην μερική απασχόληση και ο μισθός ε, ανά ώρα ε, είναι χαμηλότερος. Αυτά τα συστατικά δεδομένα λοιπόν βασίζονται σε τέτοιου είδους στοιχεία. Κάτι άλλο. Το 2005 όταν εγώ συνέταξα τη δική μου την έκθεση, η διαφορά ήταν 15%, τώρα αυτή η διαφορά έχει ανέβει στο 17%. Ε, δεν είναι η κρίση γιατί τα στοιχεία αυτά είναι του 2007. Τρίτη ερώτηση. Τι θα γίνει τελικά με τις ε, προτάσεις ε, τις οποίες καταθέσαμε εμείς στην τελευταία μας έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλετε και ένα σύντομο σχόλιο από την εκπρόσωπο της Κομισιόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Κοιτάξτε, η διαφορά ανάμεσα στο 15% που είχατε εσείς στην έκθεση σας, κυρία Μπάουρ, και το 17% είναι η διαφορά για να υπολογιστεί, ε, είναι διαφορά υπολογισμού. Διαφορά υπολογισμού έγινε και κατά τα άλλα, το τι κάνουμε για να εφαρμόσουμε τις προτάσεις σας στην πρακτική. Κοιτάξτε, δουλεύουμε πάνω σε αυτό, πήραμε κάποιες προτάσεις και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και με τις υπόλοιπες. Κατόπιν, το ερώτημα που αφορά στο γιατί δεν διαφημίσαμε και στις πέντε χώρες ε, ε, μάλλον μόνο σε πέντε χώρες και όχι σε όλες τις χώρες. Κοιτάξτε, διαφημιστήκαμε σε όλες τις εφημερίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι σε όλες τις χώρες, προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε μια γεωγραφική ισορροπία. Οι πέντε χώρες που σας ανέφερα, Εκεί κάναμε διαφήμιση ε, χρησιμοποιώντας τα δημόσια λεωφορεία. Η Ουγγαρία, η Πολωνία, το Βέλγιο, η Ισπανία Προσπαθήσαμε λοιπόν να διατηρήσουμε μια γεωγραφική ισορροπία και τα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας στην πρώτη φάση της εκστρατείας δεν αρκούσαν για να διευμιστούμε σε όλα τα κράτη-μέλη. Έπρεπε λοιπόν να κάνουμε μια επιλογή και προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό με τον πιο δίκαιο τρόπο. Στη δεύτερη φάση